Καλημέρα σας. Περιμένοντας να γίνουμε έξι τουλάχιστον τα μέλη και με τον κύριο Μπουσουτήλ να είναι στη διαδρομή, να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις που πάρθηκαν χτες στη συνάντηση των συντονιστών ε, σε ό,τι αφορά το μεγάλο ζήτημα των ε, μη αναφορών και μετά από μια αλληλογραφία μας με την Γενική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Εσωτερικών ε, Υποθέσεων. Ε, καταλήξαμε σε, ένα, σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χειριζόμαστε τις μη αναφορές. Δημιουργείται ένα φίλτρο για αυτές. Έτσι σε εμά θα έρχονται καταρχήν ε, όσες θεωρούμε ότι είναι αναφορές πραγματικά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπε θα απορρίπτονται. Θα είναι σε ένα register, σε ένα αρχείο, σε ένα πρωτόκολλο και οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να περάσουν από την κατηγορία των non-petitions στην κατηγορία των petitions. Υπάρχουν γράμματα αλληλογραφία σχετική με το ζήτημα. Το δεύτερο αφορά στις ε, ε επισκέψεις. Ε, the coordinators took note of the chair's announcement that they οι συντονιστές ε, σημείωσαν ε, τις ε, ανακοινώσεις της Πρόεδρου ότι εκκρεμεί ακόμα η απάντηση στην επιστολή που απεστάλλει στον Πρόεδρο Μπούζεκ. Γι' αυτό και ζητήθηκε να καθορίσουμε τι θα γίνει με τις προγραμματισμένες επισκέψεις, να γίνουν προτάσεις. Αποφασίστηκε να υπάρξει μια επιπλέον επίσκεψη στη Ρουμανία για τις προγραμματισμένες επισκέψεις και ζητήθηκε από τη Γραμματεία να προτείνει κατάλληλες ημερομηνίε. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι συντονιστές αποφάσισαν ότι η επίσημη πρόσκληση θα πρέπει να αποτανθεί στον Επίτροπο Ποτότσνικ ε, προκειμένου να έρθει εδώ να μιλήσει στην ε, Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα το Δεκέμβριο για να ε, συζητήσουμε τα θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εν ώψη και της προετοιμασίας μιας μελλοντικής ανακοίνωσης επί του θέματος. Όσον αφορά τώρα τις προσκλήσεις προς τους αναφέροντες και την παρουσία τους στις συνεδριάσεις μας, οι συντονιστές αποφάσισαν ότι βάσει του κανονισμού οι αναφέροντες έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ε, υπό την αίρεση της έγκρισης της Προέδρου και επίσης επανεπιβεβαίωσαν ότι είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν για τον αριθμό των αναφερόντων που θα μπορούν να είναι παρόντες σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής και ε, επίσης ότι ο χρόνος αγόρευσης των αναφερόντων ε, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Προέδρου και δεσμεύτηκαν να προσπαθούν να καθορίσουν την ημερήσια διάταξη κατά τρόπον ώστε να μπορεί να δίνεται ο λόγος στους αναφέροντες όταν είναι παρόντες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει επαρκής χρόνος για να κάνουν τις δηλώσεις τους. Οι συντονιστές αποφάσισαν επίσης ότι η συνάδελφος Σιλβάνα Κοχμερίν από την ομάδα των Φιλολευθέρων θα είναι η συγγήτρια για τη γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό του συνηγόρου του πολίτη και για το 2012 και αποφάσισαν επίσης ότι θα γίνει και μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Κάτι το οποίο όμως ε, έχει ακόμα σε κρεμότητα τα θέματα περιεχομένου και μερίσιας διάταξης. Ελήφθη επίσης μια επιστολή από τον πρόεδρο Μπούζεκ για την αμόχωστο. Υπήρχε ένα μήνυμα επίσης από τον Ισπανό Δημόσιο ε, Συνήγορο του Πολίτη, το οποίο δεν διάβασα. Όσον αφορά τώρα την αμόχωστο, μου ενημερώθηκα ότι υπάρχει, δεν ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τις επαφές με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο πρόεδρος Μπούζεκ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα της αμοχώστου. Μετά από τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά λοιπόν για τις αποφάσεις των συντονιστών. Κύριε Μποστινάρου, καλημέρα σας. Ε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Ähm, ähm, καλημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι αυτή τη φορά αντιλαμβάνουμε ότι για πρώτη φορά όσον αφορά την περίληψη και τις υποδείξεις σχετικά με τις αναφοράς θα αναφέρεται η τελική ημερομηνία προθεσμίας που μπορεί κανείς να παρέμβει κατά τρόπον ώστε να μπορεί κανείς να αναφερθεί και προφορικά σε αυτές τις αναφορές και ελπίζω ότι αυτή η πρακτική θα ισχύσει και στο μέλλον. Επίσης εγώ κατάλαβα διαφορετικά το θέμα αυτό, δηλαδή νόμιζα ότι ο διαμεσολαβητής μεσολαβητής αρνήθηκε να εμφανιστεί προς συζήτηση. Δεν ξέρω εάν δεν τον βόλευαν οι ημερομηνίε ή δεν μπορούσε ή για ποιο λόγο δεν ήρθε και θα ήθελα οι συντονιστές να ασχοληθούν με το θέμα αυτό και κάθε φορά πριν ε, ξεκινήσει μία νέα προεδρία ίσως θα ήταν καλό να ζητούμε από τον διαμεσολαβητή της χώρας να έρχεται να συζητήσει μαζί μας. Θα σας απαντήσει η γραμματεία. Έχουμε ένα αντίγραφο της απάντησης που λάβαμε από τον Ισπανό Συνήγορο του Πολίτη και έχει προσθεθεί στα έγγραφα που λαμβάνετε μαζί με την ημερήσια διάταξη. Εάν δεν το έχετε μπορώ να σας δώσω ένα αντίγραφο. Δυστυχώς είναι στα Ισπανικά. Ε, πρόεδρος, γι' αυτό άλλωστε και εγώ δεν μπορούσα να εξηγήσω περισσότερα. Μπορεί ο κύριος Μάγερ να σας δώσει κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω. Θέλετε την επιστολή του Ισπανού διαμεσολαβητή? Ωραία, θα σα δοθεί. Εγώ θα παρακαλούσα να το να αξιολογήσουμε αυτό το έγγραφο στην Επιτροπή διότι νομίζω ότι καταρχήν όλα τα μέλη της Επιτροπής είχαν εκφράσει την επιθυμία αν υπάρχουν προβλήματα σε μία χώρα να έρθουμε σε επαφή και να κάνουμε κάποιο διάλογο κατόπιν προσκλήσεως είτε με την αρμόδια Επιτροπή Αναφορών ή με τον διαμέσολαβητή, τον Ombudsman ε, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Ήταν καλό δηλαδή ε, κάποια στιγμή να συζητήσουμε με έναν διαμεσολαβητή μπορούμε και να τσακωθούμε διότι ενδέχεται ορισμένα θέματα να πρέπει να συζητηθούν και κλεισμένων των θυρών πάντως θα πρέπει να γίνει μια περαιτέρω αξιολόγηση. Ε, ε ίσως είχα αντιληφθεί λανθασμένα το θέμα διότι η υπήρχαν και άλλα, άλλες αναφορές όπου καλό θα ήταν να μπορούσαμε να καλέσουμε τον ε, ε, συνήγορο του πολίτη κατά τρόπον ώστε να συζητήσουμε μαζί του το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή και το περιεχόμενο του διαμεσολαβητή του πολίτη της Ισπανίας στην Επιτροπή. Ε, με συγχωρείτε, αλλά ε, μου μετέφρασαν ένα μέρος από την ε, ομιλία της Ισπανίδος συνηγόρου του πολίτη και είπε ότι αυτό δεν είναι στα πλαίσια της εντολής της και εφόσον το θέμα βρίσκεται στα ισπανικά δικαστήρια θα περιμένουμε. Πάντως πιστεύω δεν είναι καθόλου κακή η πρότασή σας. Εάν υπάρχουν πολλές αναφορές από μία χώρα, η επαφή με το συνήγορο του πολίτη του αρμόδιας χώρας δεν είναι καθόλου κακή και θα μπορούσαμε ίσως να καλέσουμε και ε, τον Ευρωπαίο συνήγορο του πολίτη. Δεν είδα τον κύριο Μπούσουτιλ. Μπορείτε να περιμένετε κυρία Άουκεν. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, ε, η καλή διοίκηση είναι, ε, ε, είναι καλή διαχείριση και διαφάνεια. Άρα δεν θα έπρεπε να έρθει ένα συνήγορο του πολίτη και κλεισμένων των θυρών. Καλό θα ήταν να τον καλέσουμε και να καλούμε τους εκπροσώπους των διαφόρων κρατών μελών αλλά αυτή η συνάντηση θα έπρεπε να συνάδει με τη σωστή και χρηστή διαχείριση και αν έχουμε πολλές περιπτώσεις από κάποια χώρα όπου πιστεύουμε ότι θα έπρεπε το θέμα να διεκπαιρεωθεί στην χώρα και υπάρχει κακή διαχείριση θα ήθελα απλώς να τονίσω ότι εγώ τουλάχιστον θα ζητούσα η κοινή μας συνεννόηση και συζήτηση να γίνει σε ανοιχτή συνεδρίαση όχι και κλεισμένων των θυρών εφόσον πρόκειται για κάποιον εθνικό συνήγορο του πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, στο... δεν είναι το ίδιο θέμα, αλλά ήρθα στην αρχή της Επιτροπής διότι ε, θα είμαι στη συνέχεια στις ψηφοφορίες της ε, Επιτροπής μου. Θέλω να σας μιλήσω για το Jugendamt, το Γραφείο Νέων και να ζητήσω ε, από τα από την Επιτροπή αυτή όποιος ενδιαφέρεται να έρθει στην ομάδα εργασίας διότι έχουμε αναφορές οι οποίες φτάνουν στα χέρια μας συχνά και πρέπει καταρχήν να τις κατατάξουμε κατά τρόπον ώστε να γνωρίζουμε ποιες είναι όντως αποδεκτές, παραδεκτές και ε, παρόλο που θα δείτε ότι υπάρχει δυσκολία στην κατάταξη αλλά πρέπει να καταταγούν για να μπορούμε καλύτερα να κατευθύνουμε τις ε, ε, αναφορές που θα φτάσουν στα χέρια μας. Αυτή είναι η πρώτη φάση εργασίας. Η δεύτερη είναι να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη με τους Γερμανούς συναδέλφους όσον αφορά τις μεθόδους και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι είναι δύο εθνικοτήτων με τους Γερμανούς σε περίπτωση διαζυγίου αν υπάρχουν ανισότητες, αδικίες και να βασιστούμε στην ε, γλώσσα η οποία δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά τρόπον ώστε να γίνει μετά η συγκριτική μελέτη. Όσο περισσότερα μέλη θα έχουν έχουμε στην Επιτροπή, τόσο περισσότερα στοιχεία θα μπορέσουμε να έχουμε και τόσες περισσότερες λύσεις θα μπορούμε να προτείνουμε. Θέλω λοιπόν να ε, ξανακάνω μία έκκληση για υποψηφίους για να συμμετάσχουν στην Επιτροπή που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Είναι ανοιχτή η πρόταση για όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την Επιτροπή. Κύριος Μάγερ. Εγώ θα ήθελα απλώ για να σας διευκολύνω να σας πω για τη, λίγο τη μετάφραση της επιστολής που έστειλε η Ισπανίδα συνήγορος του πολίτη. Ε, για την πρόσκληση που της έγινε για να παραστεί εδώ και να εξηγήσει τι γίνεται με την ομοθεσία για τις παράκτιες περιοχές της Ισπανίας. Η επιστολή, επειδή είναι στα ισπανικά, σα τη μεταφράζω εγώ, λέει καταρχά ότι λυπάται η συνήγορο του πολίτη που δεν μπορεί να παραστεί. Κατά δεύτερον, παραπέμπει στα όσα υπερασπίζεται και μας παραπέμπει στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο και μία σειρά από ανακοινώσεων που υπάρχουν και επίσης λέει ότι επειδή το συνταγματικό δικαστήριο ε, θεωρεί ότι ισχύει παράκτια νομοθεσία, θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να παραστεί. Αυτό λέει η επιστολή συγκεκριμένα. Λοιπόν, πρέπει να διαχωρίσουμε δύο θέματα. Το ένα είναι η ε, δήλωση ενός συνηγόρου του πολίτη ή η παράσταση ενός ε, αντιστοίχου ατόμου εδώ στην Επιτροπή και ε, φαντάζομαι ότι ο συνήγορος του πολίτη μπορεί να καταλήξει σε μία απόφαση. Αλλά στην Ισπανία όλες οι διαδικασίες δεν ήταν νομότυπες και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο μπορούμε να απευθύνουμε ή το συνήγορο του πολίτη. Δηλαδή να δούμε ε, αν σε περίπτωση αναφορών που αναφέρονται σε νομικά θέματα ε, πρέπει να τα παραπέμπει εις το Λουξεμβούργο στο αρμόδιο δικαστήριο ή αν μπορεί ο ίδιος να τα διεκπαιρεώσει. Είναι που πρέπει να συζητήσουμε και ίσως θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή για μελλοντικές διαθεσμικές συμφωνίες να λάβουμε υπόψη μας το θέμα αυτό διότι ε, το Συμβούλιο θα πρέπει να δεσμευτεί δηλαδή να μπορούμε να απαιτήσουμε ε, από τα κράτη-μέλη ότι οι αρμόδιοι συνήγοροι του πολίτη σε εθνικό επίπεδο θα έρχονται συνεδριάσεις μας. Ε, το ίδιο είναι ε, αυτό το οποίο κάνουμε όταν συζητάμε με υπουργού ε, πριν την ανάληψη μιας προεδρίας. Να τους ζητάμε δηλαδή να προσέλθουν ένα-δύο μήνες πριν αναλάβουν την προεδρία και ε, συγχρόνως ο συνήγορος του πολίτη, του κοινοβουλίου, της αρμοδίας χώρας που θα αναλάβει την προεδρία να έρθει κατά τρόπον ώστε να έχουμε μία τέτοια δημόσια ανταλλαγή απόψεων ε, αν ε, θέλουμε να ακούσουμε όμως μία αξιολόγηση ενός ε, συναδέλφου ο οποίος θα μας πει θα σας πω περισσότερα εάν είμαστε κεκλεισμένοι των θυρών θα το ξανασκεφτούμε διαφορετικά θα πρέπει οι συνεδριάσεις να είναι δημόσιες και οι συνήγοροι του πολίτη και οι υπουργοί θα πρέπει να προσέρχονται ακόμη και αν έχουμε λεπτά θέματα προς συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών θα ήθελα λοιπόν να ξέρω και τις άλλες απόψεις. Έχω σοκαριστεί λίγο ε, για την αντίδραση του Ισπανού διαμεσολαβητή. Μιλάει ως Σαν να έχει αναθέσει θέματα και δεν μπορεί να βρίσκεται αυτός εκεί. Ας έρθει εδώ να μας εξηγήσει και να μας πει. Μερικές φορές ε, έχουν πρόβλημα με τον ε, διαμεσολαβητή στην Ισπανία, τότε συνειδητοποίησα και πριν. Ε, και όχι μόνο στη Δανία αλλά και σε άλλα μέρη και ε, πελείτομε με αυτή την απάντηση. Δεν είναι τρόπος να συμπεριφέρεται κανείς ο συνήγορος του πολίτη. Αντιπροσωπεύει τον λαό και θα πρέπει να είναι η φωνή του πολίτη. Πραγματικά μένω έκπληκτη. Uh, Να το συζητήσουμε ως μέρος της επόμενης συνάντησης. Να συγκεκρινοποιήσουμε λίγο την θέση μας απέναντι, γενικώ απέναντι στους συνηγούρους του πολίτη. Ας το αφήσουμε για την επόμενη συνέδρια. Σας ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Η αναφορά του κυρίου Σάντρο Μίτσι από την Μάλτα εξ ονόματος της Harpoon Fishing Association σχετικά με τις άδειες αλληλείας που διατίθενται στη Μάλτα. Ε, we do not have any petitioner. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Εκ μέρους της Κομισιόν η κυρία Σκάλκο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσει τον αναφέροντα που ήγηρε αυτό το θέμα που σχετίζεται με την συμμόρφωση με τον κανονισμό 1967 του 2006, την λεγόμενη, το λεγόμενο κανονισμό για τη Μεσόγειο. Όπως, αναφέρεται στην απάντηση της Κομισιόν, οι πρακτικές που ασκούσε ο ε, αναφέροντας ε, απαγορεύοντας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του κανονισμού. Αυτός ο κανονισμός ε, έχει τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2007 και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Ε, δεν προβλέπεται παρέκκληση στην χρήση ψαροντούφεκων με μπουκάλα οξυγόνου και αυτό διασφαλίζει μια ισότιμη μεταχείριση για όλους τους αλληλείς στις χώρες της Μεσογείου. Θέλω να τονίσω ότι μετά τη δεύτερη ανακοίνωση από τον αναφέροντα η ε- Κομισιόν επικοινώνησε με τις αρχές στην Κύπρο διότι ο αναφέροντας ισχυριζόταν ότι στην Κύπρο ξέδιδαν άδειε αλίας για την αλία με χρήση ψαροτούφεκων και επικοινωνήσαμε με την Κύπρο να δούμε αν η απαγόρευση είχε ε, τεθεί σε εφαρμογή στην Κύπρο και μα έχουν επιβεβαιώσει ότι από την θέση ισχύ της, ε, του κανονισμού του Μεσογειακού η οδηγία αυτή δεν, μάλλον οι αρχές δεν έχουν, ακόμη, δεν έχουν πια εκδώσει άδειε διότι δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Μας έχουν δώσει και κάποια στοιχεία σχετικά με τις παραβιάσεις, σχετικά με την χρήση ψαροτούφεκων το 2010 στην Κύπρο και τον αριθμό αυτών των παραβιάσεων που σχετίζεται με τη χρήση ψαροτούφεκων σε σχέση με μπουκάλα οξυγόνου. Η Κομισιόν δεν έχει στοιχεία ε, μη εφαρμογής της απαγόρευσης στην Κύπρο. Αυτή είναι η απάντησή μας στον αναφέροντα. Thank you, Madam Chair. Uh, Ο κύριος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και την εξήγηση που μας έδωσε. Δύο σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Το πρώτο αφορά την αλία με ψαρωτήφεκο σε μία άλλη χώρα, την Κύπρο. Ο αναφέρον έκανε προσωπική έρευνα επί του θέματος και διαπίστωσε ότι υπάρχουν άδειες ε, στην Κύπρο και δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι διαθέσιμε σε μια άλλη χώρα, αλλά το γεγονός ότι του απαγορεύεται να ασκήσει αυτή τη μορφή αλίας στη χώρα του. Η Επιτροπή μας επιβεβαίωσε δύο πράγματα. Ότι αυτό φαίνεται ότι είναι σαφώς απαγορευμένο βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αυτό το δέχομαι γιατί είναι σαφή ο νόμο. Και το δεύτερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις Κυπριακές Αρχές και επιβεβαίωσαν ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν επιτρέπεται πλέον. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στον αναφέροντα ο συγκεκριμένος άνθρωπος διαπίστωσε ξαφνικά ότι η επιβίωσή του, διότι η επιβίωσή του είναι αυτή που έχει σημασία, είναι πλέον παράνομη ε, βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τον Ιούνιο του 2007. Είναι πολύ εύκολο να καθόμαστε εμείς στις καρέκλες μας στις Βρυξέλλες και να λέμε αυτό είναι παράνομο, τελεία και παύλα. Φανταστείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οικογένεια, ο οποίος έχει ένα τρόπο να εξοικονομεί τα προστοζήν και ξαφνικά από τον Ιανουάριο του 2007 κάποιος του λέει ξέχνατο, δεν μπορείς πλέον να βγάζεις ε, το ψωμί σου με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να δεις ε, πώς μπορείς να επιβιώσεις με άλλο τρόπο. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει και, αυτό το, και αυτή την πτυχή της ε, νομοθεσίας. Δεν μπορούμε να λέμε απλώς ότι απαγορεύεται η αλία ψαρετούφεκου με μπουκάλα οξυγόνου και τελείωσε το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζήτησε να έχουμε ένα ισότιμο πεδίο. Πραγματικά θα ήθελα να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι στους όρους έχουμε όταν ένας άνθρωπος απαγορεύεται να ε, ψαρέψει με ψαροντίφεκο, με μπουκάλα μόνος του. Ε, και τι γίνεται όταν έχουμε ψαρότρατες που αλλιεύουν σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό όμω το οποίο θα ήθελα να μου απαντήσει κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εξής. Τι εναλλακτική λύση προτείνεται σε ανθρώπους, ε, σε μια κοινότητα ανθρώπων που ξαφνικά καταστράφηκε ο βασικός ε, βιοποριστικός τους ε, πόρος. Και θα πρέπει λοιπόν να τους δοθεί μια εναλλακτική λύση. Δεν μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος αλλιεύει ε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ε, είτε μας αρέσει είτε όχι, ε, αλλά αυτός εξοικονομεί τα προστοζήν με αυτόν τον τρόπο και να έρθουμε ξαφνικά το 2007 και να του πούμε ότι απαγορεύεται πλέον να ασκεί το επαγγελμάτο. Πρέπει να του δώσουμε μια εναλλακτική λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια εναλλακτική λύση και να εξηγήσει στη συγκεκριμένη κοινότητα λιέων ότι μπορούν να ε, κάνουν κάτι άλλο και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τον βοηθήσει να κάνει κάτι άλλο. Πραγματικά θα ήθελα μια εξήγηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τι ανησυχίες που μόλι σα εξέφρασα. Ευχαριστώ. We had Έγινε μια συζήτηση ανάμεσα στους συντονιστές ε, για το πώς ε, θα δίναμε επαρκή χρόνο και να μην έχουμε πράγματα στην μερίσια διάταξη που να μην ε, αξίζει να ταπανούμε χρόνο για αυτά. Θα το δούμε ξανά και ξανά. Τι γίνεται με την αλία των φαλενών. γιατί και εκεί εμείς καθόμαστε και κάθεται και η Επιτροπή και προσπαθούμε να δούμε πώς ένας αλλιές μπορεί να βρει ένα άλλο τρόπο, μια άλλη μέθοδο αλλιείας. Ε, ζητών από την Πρόεδρο να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια. Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο να ζητήσουμε από την Κομισιόν να σπαταλήσει περισσότερο χρόνο για να μας εξηγήσει για κάτι για το οποίο δεν είναι αρμόδιο είναι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που κάνουν τους νόμους. Έχουμε ε, κάνει αυτό το νόμο, είναι σαφής και μπορεί να βρεθεί μια άλλη αλλιευτική μέθοδος. Νομίζω είναι χάσιμο χρόνο να καθόμαστε και να κάνουμε αυτή τη ζήτηση εδώ. Πραγματικά υποσκάπτουμε όλων των ειδών της νομοθεσίας αν κάθε φορά ε, αναζητούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει κανείς αν αυτό δεν είναι νόμιμο. Ελάτε τώρα. Ευχαριστώ. πραγματικά διαφωνώ. Δεν είναι χάσιμο χρόνο. Θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Ε, ακριβώς αυτό είπατε. Ακριβώς αυτό είπατε. Όταν κάποιος υποβάλλει μια αναφορά και όταν το προς τον ζήνα αυτού του ανθρώπου και της οικογένειάς του διακυβεύονται, το, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να του δώσουμε μια απάντηση. Η απάντηση μπορεί να είναι αυτή που δεν θέλει να ακούσει ο αναφέρον. Αλλά έχουμε καθήκον να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το άτομο και στην οικογένειά του. Και δεν πρέπει να πούμε ότι είναι χάσιμο χρόνου. Πραγματικά επιμένω να πάρουμε μια απάντηση από την Κομισιόν ως προς το ποια εναλλακτική λύση προτείνει η Κομισιόν για αυτό το άτομο του οποίου έχει σταματήσει η διαβίωσή του και τα προσωρινή του με αυτόν τον τρόπο. Α, ah, yes, Äh, Πιστεύω ότι το ουσιαστικό πρόβλημα ε, και ο συνάδελφος Μουσουτήλ έχει δίκιο. Πάντοτε υπάρχουν αλλαγές, ιδίω στο γεωργικό τομέα, ε, το ε, έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένως. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί για τους ενδιαφερομένους από πλευράς του διαφερομένου και έχουμε κάνει τέτοιες έρευνες αλλά αυτό το οποίο προσέχουμε συνήθως και ο στόχος μας είναι να μπορέσουν να συμμετέχουν και οι ενδιαφερόμενοι γι' αυτό και έχουμε προθεσμίες γι' αυτό ζητούμε οι γεωργοί ή οι οικογένειές τους να έχουν τη δυνατότητα να καταρτήσουν μια εναλλακτική λύση και αυτό το οποίο λυπάται ο κύριος Μπουσουτήλ δεν είναι η απαγόρευση αλλά πλούστατα ότι ξέχασαν να, να πούν στα άτομα αυτά πώς θα πάνε από το σημείο α στο σημείο β, πώς θα αλλάξουν τη ζωή τους. Και από αυτού έχει δίκιο. Τώρα, εάν είναι κάτι που πρέπει να αναλάβει η Επιτροπή, είναι διαφορετικό, διότι όπως είπε η κυρία Άουκεν, υπάρχει μία νομοθεσία στην οποία συμμετείχε το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, άρα υπάρχουν πολλοί συνυπεύθυνοι. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει ε, ίσως να έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή η οποία κατήρτισε αυτή την νομοθεσία να τους παραπέμψουμε το έγγραφο αυτό και να τους πούμε δέστε πού καταλήξαμε τώρα για να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ των Βρυξελών και προφανώς με το κράτος μέλος, γιατί συμμετέχει και το κράτος μέλος η Μάλτα. Δεν είναι στο κενό δηλαδή αυτή η διαδικασία. Θα έλεγα λοιπόν να αφήσουμε αυτή την αναφορά ανοιχτή, να κοιτάξουμε ποια ήταν η αρμόδια επιτροπή και να τους ζητήσουμε να ασχοληθούν συγκεκριμένα με το θέμα, διότι ένα πράγμα είναι η απαγόρευση και άλλο είναι να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις στους ενδιαφερόμενους και πληττόμενους και αυτό ακριβώς δεν λήφθηκε υπόψη και είναι θέμα ε, αποδοχής ε, ακριβώς εκεί που τίθεται το πρόβλημα. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε να ε, γίνει αποδεκτό, διότι αν δεν έγινε αποδεκτό σημαίνει ότι δεν έγινε καταληπτό και τρίτον το πιο δύσκολο είναι ότι ενδεχομένως η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί παράνομα και αυτό απευχόμαστε γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Αρμόδια Επιτροπή να καταρτήσει μια σχετική γνωμοδότηση. Πράγμα έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το νομικό, το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δεν μπορούμε ξαφνικά να αμφισβητούμε με μια συγκεκριμένη περίπτωση την νομοθεσία την οποία έχουμε εγκρίνει και ως, ε, ως ευρωβουλευτές και εδώ έχει η κυρία Άουκεν δίκιο. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν μπορούμε να επανέρθουμε σε μια περίπτωση η οποία ε, μπορεί να μην είναι ατομική και να έχει περισσότερους, ε, να έχει επιπτώσει σε περισσότερο αριθμό, σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Θα έλεγα λοιπόν ότι μία, ε, η πρόταση του κυρίου Γιάρ να ζητήσουμε από την, από την Κομισιόν μία, από την, Επιτροπή για τα ψάρια, για την αλία ε, μία, μία, μία εναλλακτική όπως τη λέτε εσείς δεν θα ήταν άσχημο ε, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι ακυρώνουμε την νομοθεσία που ήδη έχουμε ε, ψηφίσει. Ε, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή και δεν ξέρω αν η κυρία Σκάλκο θα ήθελε από την Επιτροπή να απαντήσει στο συγκεκριμένο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα αξιότιμα μέλη για τα σχόλιά τους. Συμφωνώ με την ανάλυση σας. Ε, το γεγονός είναι όμως ότι εδώ έχουμε δύο θέματα. Αφενός ε, υπάρχει ο αναφέρον που λέει ότι υπάρχει αντίστοιχη πρακτική στην Κύπρο και επομένως ε, Εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι εκδίδονται άδειες ε, και οι Κύπροι αλληλείς έχουν στην κατοχή τους άδειες για τη διεξαδογή της συγκεκριμένη δραστηριότητες, θα θέλαμε να τους ζητήσουμε ε, να ξεκινήσει καταγγελία επί του θέματος. Από πλευράς ε, ελέγχων τώρα, ο έλεγχος είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρκετά μέσα για να εξετάζει ότι συμμορφούνται προς τους κανόνες τα κράτη-μέλη και θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά για να διασφαλίσουμε ότι γίνεται σωστή εφαρμογή. Όσον αφορά τώρα τις εναλλακτικέ. Υπάρχει κοινωνική και οικονομική ανησυχία των επιπτώσεων συγκεκριμένη ε, διάταξης ε, για τη διαβίωση αυτών των ανθρώπων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται με αυτή την ανησυχία, αλλά θα ήθελα να πω ότι ο κανονισμός αυτός αφορά πάρα πολλές πτυχές της αλίας και κυρίως αλλιευτικές πρακτικές οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους αλλιευτικούς πεόρους και το περιβάλλον. Για παράδειγμα, για τις τραέτες που αναφέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στον κανονισμό αυτό. Δεν ε, ασχολόμαστε μόνο με τις πρακτικές αλλία με ψαροτούφακο που κάνουν ε, ερασιτέχνες αλλιείς ε, ή οργανώσεις αλλιέων, αλλά και με άλλες πρακτικές. Πρόκειται για ένα συνολικό κανονισμό που έχει πάρα πολλές διατάξεις και πολλούς περιορισμούς που ισχύουν για για τις και για τις μεγαλύτερες αλληλευτικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τις εναλλακτικέ, ε, να σας πω ότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, το οποίο ε, δίνει και χρηματοδότηση για αλλαγή αλληλευτικών δραστηριοτήτων και εδώ είναι ευθύνη τη αρμόδια αρχή του κράτους μέλους να αναθέσει συγκεκριμένα κονδύλιο. Ίσως λοιπόν ο αναφέρον θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες εθνικέ αρχές για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλαία για να δει τι δυνατότητες έχει να αλλάξει τη δραστηριότητά του η οποία δραστηριότητα βάσει του κανονισμού για τη Μεσόγειο εξακολουθεί να είναι παράνομη. Μικρόφωνο παρακαλώ. Anything to be added to this explanation? Θέλετε να προσθέσετε κάτι, είστε ικανοποιημένος κύριε, κύριε Μπουσούτηρ. Ναι, είμαι ικανοποιημένο για το πρώτο σημείο, δηλαδή αυτό το άτομο φυσικά δεν γνώριζε ότι απαγορευόταν αυτή η μέθοδος μέχρι να τον σταματήσουν, διότι οι φίλοι του στην Κύπρο εξακολουθούσαν να την κάνουν. Τώρα είναι σαφές ότι δεν είναι παράνομο μόνο σε μια χώρα, αλλά και στην άλλη. Αυτό είναι σαφές. Το δεύτερο είναι λιγότερο σαφές όμως. Ως Επιτροπή θα πρέπει να το απαντήσουμε και να πούμε ότι θα πρέπει να του δώσουμε μάλλον πληροφορίες ως προς τις εναλλακτικές λύσεις που παρέχονται για αυτόν, διότι είναι σοβαρό. Θα πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να ε, ζήσει και ε, η βοήθεια της Κομισιόν θα ήταν πολύ χρήσιμη. Αντί να πάμε στην Επιτροπή Αλίας, να του δώσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για το πού πρέπει να απευθυνθεί για να βρει βοήθεια για να ξαναξεκινήσει τη ζωή του, διότι περί αυτού πρόκειται. Δεν ε, υπάρχει αμφιβολία ότι ποτέ δεν είχα ζητήσει την απαγόρευση ή τη μη τήρηση της νομοθεσίας. Αυτό που λέω είναι ότι αν ο νόμος σταματάει μια πρακτική που επηρεάζει ε, τη μια οικογένεια, θα πρέπει να σκεφτούμε τι εναλλακτικέ λύσει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τους δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μπουσουτήλ έχει δίκιο, αλλά εγώ θα ήθελα να το διευρύνουμε. Δηλαδή θα έπρεπε να παραπέμψουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Αλληλείας. Νομίζω ότι θα ήταν λογικό, διότι ε, ε, δεν, ε, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει η Επιτροπή Αλληλείας να ασχοληθεί και με τις εναλλακτικέ λύσεις για την εξέβρεση εισοδήματος. Νομίζω ότι δεν χάνουμε χρόνο εάν εξετάσουμε και τις δύο εναλλακτικές εναλλακτικέ. Δηλαδή και να παραπέμψουμε στην Επιτροπή Αλίας όπου το θέμα συζητιέται, αλλά θα, καλό θα ήταν να σκεφτούν οι εμπειρογνώμονες και τις ε, εναλλακτικέ με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τρόπο ώστε να έχουμε ε, ε, απαντήσεις. Δεν χρειαζόμαστε ατελείωτο χρόνο, δηλαδή νομίζω ότι μια παράλληλη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, της Επιτροπής Αλληλείας θα μπορούσαν ε, να επιταχύνουν για να υπάρξει μία απάντηση στον ενδιαφερόμενο διότι στο τέλος θα χρειαστεί να εμπλακεί και η Μάλτα. Δηλαδή αφού αποφασίσουν οι επιτροπές θα, θα πρέπει επιτροπού το κράτος ε, να συμπράξει για να δει πώς θα εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο η απόφαση στον αναφέροντα αφού έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες παράλληλα όμως και με τη διαβεβαίωση της Επιτροπής ότι στην Κύπρο τυπικά με βάση ό,τι στοιχεία έχουμε δεν ισχύει κάτι τέτοιο ή αν ισχύει. Ακούσαμε ότι στην Κύπρο δεν ισχύει με βάση τις επαφές που είχε η Επιτροπή. Ε, επομένως το θέμα έχει και την άλλη διάσταση. Και αυτό πρέπει να το ε, λάβουμε υπόψη. Άλλωστε να μην ξεχνούμε ότι κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει επίσης ερώτηση προς την Επιτροπή. Και αναρωτιέμαι αν κύριε Μπουσουτήλη, εσείς ή κύριε και ή κύριος Γιάρ ή και εγώ θα μπορούσαμε ως μέλη του Κοινοβουλίου να υποβάλουμε μια τέτοια ερώτηση προς την Επιτροπή ε, και να δούμε τι μπορεί να μας απαντήσει. Ενώ την ε, Επιτροπή Αλίας στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σαν Αυστριακή βεβαίως δεν είμαι ειδική στην αλληλεία αλλά υπάρχει και ένα θέμα. Είναι ένας μόνος αναφέρον ο οποίος πλήττεται από αυτό το πρόβλημα ή είναι περισσότεροι γιατί είναι μία άποψη η οποία θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Δεν είμαι εμπειρογνώμων, δεν θέλω να επισέλθω σε μία ειδική συζήτηση αλλά εδώ μιλάμε για τη μοίρα μίας οικογενείας ή πρέπει να δούμε ε, πώς θα άτομα έχουν ε, πληγεί από αυτή την νομοθεσία. this in my suggestion. Το είχα αναφέρει και εγώ στην πρότασή μου. Ε, εντάξει, κρατούμε ακόμα ανοιχτό, ανοιχτή την αναφορά. Παρακαλώ κύριε Μπουσιτέλ, ναι, επειδή η συνάδελφος ε, ενδιαφέρθηκε, θα πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για μια μικρή κοινότητα ανθρώπων, πολύ μικρή, και είναι απλώς ε, αλία με ψαροντούφεκο, βουτάς με μπουκάλες και αλιεύεις ψάρια και έτσι εξοικονομείς τα προστοζήν. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μικρή κοινότητα, 50 άτομα το πολύ, τουλάχιστον για τη χώρα μου. Ε, φαντάζομαι ότι αντίστοιχο αριθμό ε, τέτοιων αλλιών έχουμε και στην Κύπρο. Επειδή όμως είναι μικρός αριθμό αριθμός δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουν τη δέουσα προσοχή όταν ξαφνικά τους απαγορεύεται το βασικό βιοποριστικό τους μέσο. Τους ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον σας. Λοιπόν, την κρατούμε ανοιχτή, περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες και τα ξαναλέμε. <clears throat> Πάμε στην ε, αναφορά 980 του 2007 του κυρίου Τόρκιλντ Ντότζεν, δανεικής καταγωγής, εξ ονόματος της ομάδας πολιτών, σχετικά με το σχέδιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου ανάμεσα στο Κίπλεφ και στο Ζόντερμπορκ στη Δανία. Ο αναφέρον έχει έρθει. Μπορεί να πάρει το λόγο. Πού να αναφέρω. Okay.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 Σήμερα έχω έρθει σαν πολίτης εδώ για να σας πω περί τίνος πρόκειται και τι σημαίνει αυτό το σχέδιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου διότι ε, πρόκειται να καταστραφεί ένας χώρος ο οποίος προστατεύεται από την Natura 2000. και ο αυτοκινητόδρομος αυτός απαιτεί η περιοχή αυτή να γίνει ένας θύλακας μεταφοράς και θα κατακαιρματιστεί επιπλέον λόγω της ε, συγκοινωνίας η οποία θα ενταθεί στο υπάρχον σύστημα αυτοκινητοδρόμων. Επιπλέον θα υπάρξει επιβάρυνση από το διοξίδιο του άνθρακο των αυτοκινήτων. Ε, θα μπορεί ίσως ε, να χτυπήσουν και τα ζώα τα οποία θα περνούν από εκεί και θα είναι μία θανάσιμη παγίδα για τους πολίτες οι οποίοι δεν θα μπορούν να περάσουν από αυτό τον αυτοκινητόδρομο εις ε, το ε, άρθρο 6 παράγραφο 3 ε, έχει προστατευθεί προστατεύεται ο χώρος Natura 2000 και εσκεμένα παρέβλεψαν αυτές τις διατάξεις οι ενδιαφερόμενοι. Βλέπουμε ότι η περιοχή αυτή διέρχεται από την περιοχή Natura 2000 και ε, υπάρχει και ε, ο αυτοκινητόδρομος του Φλένσμπουργκ που διαπερνά αυτή την περιοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο οι αλλαγές ε, ε, για το σύστημα αυτοκινητοδρόμων και για το δίκτυο θα επιφέρουν αλλαγές και για το προστατευόμενο χώρο αυτό και θα συσσωρευτούν περισσότερες επιβαρύνσεις οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί ε, αν υπάρξουν, υπάρξει χρησιμοποίηση αποδομικά υλικά για να σταθεροποιηθεί το υπέδαφος του αυτοκινητοδρόμου. Θα δημιουργηθεί σκόνη η οποία θα επεκταθεί χιλιόμετρα πέραν του εργοταξίου και θα μπορέσει να επιβαρύνει ένα πολύ μεγάλο χώρο. Ε, δεν θα μπορεί κανείς ε, να φυτέψει τίποτα, δηλαδή υπάρχουν πολύ καλύτερες λύσεις από αυτή την οποία επιζητούν να εφαρμόσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλωστε δεν, χρειάζεται ένας τέτοιος μεγάλος αυτοκινητόδρομος για να παρακάμψει κανείς το, και να διεκπαιρεώσει τη μεταφορά από ένα μικρό νησάκι όπου υπάρχουν πολύ λίγα αυτοκίνητα. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχει παραπληροφορηθεί ε, απλούστατα για να αποφευχθεί η δικαστική ε, διαδικασία. Δηλαδή στην αιτιολόγηση ελέγχθη ότι ε, δεν υπάρχει ο χώρος αυτός Natura 2000 ε, και ε, ότι οι αλλαγές αυτές προχώρησαν όταν ήδη είχε προχωρήσει το εργοτάξιο και θα έπρεπε να υπάρξει μία επέμβαση και να διορθωθούν όλα αυτά τα λάθη. Ευχαριστώ πολύ. Όπως γνωρίζει η Επιτροπή αυτή, είναι δύσκολο να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις οικονομικές δραστηριότητες και την προστασία της φύσης, ιδιαίτερα όταν ε, έχουμε να κάνουμε το ε, Natura 2000 και χώρους ε, Natura 2000. Η ύπαρξη όμως ενός τέτοιου χώρου δεν αποκλεί εντελώ τι οικονομικές δραστηριότητες. Ο καλύτερη και η χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτή είναι να γίνει μία αξιολόγηση των επιπτώσεων. Και αυτό που κάνανε οι Δανέζικες αρχές, ε, κάνανε μία ανάλυση των ε, επιπτώσεων στον δρόμο. Χάρη στην αναφορά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την ποιότητα των αξιολογήσεων αντικτύπου και είναι γι' αυτό που η Κομισιόν ξεκίνησε μία διαδικασία με μία επίσημη επιστολή το 2008. Η αμφιβολία έγινε στην, αντίκτυπο στις θρεπτικές ουσίες, στα υπόγεια και στα πτηνά. Τώρα, στην απάντησή τους ε, στην επίσημη προειδοποίηση, οι δανέζικες αρχές υπέδειξαν ότι θα άλλαζαν ορισμένα πράγματα του προγράμματος και θα αντικαθίστατο η σύραγγα με γέφυρα. Ε, για τα στρεπτικές ουσίες έδωσαν πληροφορίες ότι το πρόβλημα δεν υφίστατο. Αναγνώρισαν το γεγονός ότι θα υπήρχε πρόβλημα για τα βατράχια και το σχέδιο δράσης ε, όπου υπάρχει αναφορά στην απάντησή μας ε, είναι δημοσίως ε, διαθέσιμο και δημιούργησαν κάποια περάσματα για τα βατράχια, γούρνες και για τα πτηνά υπέβαλαν μια μελέτη που έδειχνε ότι ο αναμενόμενος θόρυβος δεν θα προκαλούσε προβλήματα. Με βάση αυτές τις πληροφορίες λοιπόν ε, στην απάντηση που δόθηκε στην επίσημη προειδοποίηση η Κομισιόν συμπέρανε ότι δεν είχαμε αρκετά στοιχεία για να συνεχίσουμε την υπόθεση και συνεπώς η Κομισιόν αποφάσισε το Μάρτιο του 2009 να κλείσει την υπόθεση επί παραβάση. Άκουσα αυτά που είπε αναφέροντας ότι είναι απογοητευμένοι. Ε, δεν έχουμε υποδείξεις για αυτά. Ε, βέβαια μπορεί να μας δώσει τα στοιχεία αλλά η δική μας ε, επίσημη προειδοποίηση είναι δημόσιο έγγραφο. Η απάντηση από τις Δανέζικες Άρχες είναι δημοσίως ε, διαθέσιμη, μπορεί να την ε, συμβουλευτεί κανείς. Αν δεν έχουμε στεναρά στοιχεία ότι υπάρχει υπόθεση, η απόφαση της Κομισιόν να περατώσει την υπόθεση του 2009 υφίσταται. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μέχρι στιγμής τα θέματα αυτά έχουν μείνει ανοιχτά ε, διότι οι κανόνες σχετικά με την οδηγία Natura 2000 ε, απαιτούν να εξετάσουμε αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και βεβαίως πρόκειται εδώ και οικονομικές δραστηριότητες πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε αν μπορούμε να αποφύγουμε την επιβάρυνση των περιοχών Natura 2000 και πρόκειται και για τη συσσόρευση επιβαρύνσεων. Έχουμε πολλές ε, τέτοιες περιπτώσεις. Αντιλαμβάνουμε τι εννοεί ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είναι δυνατόν το κράτος να λέει δεν υπάρχουν συσσωρευτικά αποτελέσματα και δεν έχει σημασία η περιοχή Natura 2000. Ε, μπορούμε τότε να επικεντρωθούμε και στο βασικότερο, το οποίο είναι ο θόρυβος. Ή αυτοί θεωρούν πιο βασικό το θόρυβο από όλα τα άλλα ε, νομίζω όμως ότι θα θυμάστε την έκθεση που είχα κάνει για την εφαρμογή του προγράμματος Natura 2000 στα διάφορα κράτη-μέλη όπου διεφάνει σαφώς και το είχαμε συζητήσει σε αυτή την Επιτροπή πριν από δύο χρόνια. Εκεί λέγαμε ότι ακριβώς αυτά είναι ε, τα προβλήματα. Πρέπει να ελέγξει κανείς τη συσσωρευτική επιβάρυνση των διαφόρων ε, επιμέρους επιβαρύνσεων και ε, ίσως υπάρχουν, υπάρχει και εδώ το ίδιο πρόβλημα. Δεν ε, εξέτασαν αυτές τις παραμέτρους, μπορούσε να έχει γίνει κάπου αλλού αυτοκινητόδρομος και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχτεί ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει να μεταθέσει κάπου αλλού ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει απασχόληση. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν συσσωρευτικές επιβαρύνσεις και να ζητήσουμε από το δανεικό κράτος να μας αποδείξει κατά πόσον ήλεγξε τις εναλλακτικέ λύσεις και γιατί δεν τις ε, συμπεριέλαβε στους υπολογισμούς. Νομίζω αυτή είναι η μέθοδος με την οποία θα έπρεπε να προχωρήσουμε διότι ε, άλλες ε, λύσεις δεν αποτελούν εναλλακτικές οδούς. Νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε προβλήματα <clears throat> τα οποία ουσιαστικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Καλό θα ήταν να υπάρχουν επιτροπές οι οποίες θα μπορούσαν να προβούν σε μια τελείως αντικειμενική αξιολόγηση των περιπτώσεων αλλά φαντάζομαι ότι ε, ο αναφέρον θα λάβει μια επίσημη απάντηση του δανεικού κράτους σχετικά με την συλλογή στοιχείων, μετρήσεων και ούτω καθεξής. Οπότε Περιμένετε κυρία Έουκεν και άλλα στοιχεία Νομίζω ότι, ε, με συγχωρείτε που μιλάω αγγλικά, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζητά, ε, ε, τις, δεν θέτει τις σωστές ερωτήσεις και εντάξει δεν απαγορεύεται να υπάρξουν οικονομικές δραστηριότητες αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις συσσωρευτικές επιπτώσεις και τις χρήσιμες εναλλακτικές λύσεις. Πράγμα το οποίο έγινε και στην Πολωνία όπου υπήρχε ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο τελικά κατέληξε στη διατήρηση και της φύσεως. Αλλά πρέπει να εμπλακούν οι εθνικές και οι περιφερειακές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία τα καταπίνει όλα ότι δεν μας αφορά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πρέπει να επανέλθουμε να προσεγγίσουμε το δανεικό κράτος και να τους ζητήσουμε να συμπεριλάβουν στους υπολογισμούς τους τα, ε, τα συσσωρευτικά αποτελέσματα για τα λοιπάσματα για ολόκληρη την περιοχή η οποία θα πληγεί. Ε, ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι λαμβάνουμε πολλές περιπτώσεις και αυτή είναι μία εξ αυτών όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια συμβατότητα μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Εμείς εδώ σε Επιτροπή πάντα υποστηρίζουμε ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι βιώσιμη ανάπτυξη, αλλιώς δεν είναι ανάπτυξη. Και εγώ συμμερίζομαι τα όσα είπε η κυρία Άουκεν πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε επί του ζητήματος. Καταρχάς ε, να υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ οδοί και οποιαδήποτε εναλλακτική οδός θα πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Θεωρώ ότι η αρχή της βιωσιμότητας ε, θα πρέπει να ισχύει για κάθε μία από τις αναφορές που λαμβάνουμε εδώ. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αμφιβολίες για την ποιότητα της μελέτης αντικτύπου που έγινε το 2008 και έτσι έγιναν αλλαγέ από τη Δανία, νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ακολουθώντας την άγουσα που μας ε, πρότεινε η κυρία Άουκεν.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 Ε, μπορώ να σας πω ότι δεν έχουν γίνει επαρκείς ε, αξιολογήσεις σχετικά με το νέο αυτοκινικό δρομό ο οποίος θα προσφέρει έσοδα ε, και κατά αυτόν τον τρόπο όμως όσοι πηγαίνουν στο Φλένσμπουργκ θα περνούν μέσω από την περιοχή αυτή Νατούρα. Γνωρίζω τα τελευταία στοιχεία αλλά αυτό το οποίο έχει απαντηθεί σχετικά με την ερώτησή μου και την αναφορά μου δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Κύριε... Ε, μικρόφωνο. We go to the report... Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Μαρία Χωσέ Τσάβες Ρέγες που θα διασχίζει το πάρκο Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας Σιέρα Ντερακένα στη Χουέλβα. Ε, και υπάρχει και μια ε, παρόμοια ακριβώς ε, πάλι από την Ισπανία για τον ίδιο δρόμο σε μια κοντινή περιοχή αν καταλαβαίνω κανά στο πάρκο Υπήκος Διαρότσε πάλι στη Χουέλβα. Από τη μεριά της Επιτροπής ο κύριος Λουρέντσο Φάρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, μας εξήγησε η Επιτροπή, όπως εξήγησε η Επιτροπή στην ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2010 και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, η διαδικασία της αξιολόγησης αντικτύπου συνεχίζεται για αυτή την υποδομή Επίσης γνωρίζετε ότι πριν από αυτή την αναφορά η Επιτροπή είχε ξεκινήσει ένα νέο πιλότο για να διερευνήσει πληροφορίες που παρήχαν μέσω γραπτής ε, ερώτηση 4116 του 2009 από το μέλος του Κοινοβουλίου Jean Lambert και αυτός ο πιλότο αφορούσε τρει διαφορετικές οδικές υποδομές ε, που προβλεπόντουσαν με αντίκτυπο στον ίδιο χώρο, Σιέρα Ντερασένα και Πίκος τη κενδίνου συνεχίζονταν. Η απάντηση που πήραμε από τις Ισπανικές Αρχές ήταν ότι οι μελέτη αξιολόγησης κινδύνου συνεχιζόντουσαν. Η Επιτροπή έκλεισε το πιλότο, αλλά θα το παρακολουθήσουμε με τις αρχές, θα δώσουμε συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία και η επόμενη, το επόμενο στάδιο είναι να περιμένουμε τα αποτελέσματα των μελετών ε, αξιολόγησης αντικτύπου και να δούμε ιδιαίτερα ε, τον αντίκτυπο στις κοινότητες και την συμμόρφωση με τις, την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την θέματα φύσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, πρόκειται για μία οδό η οποία θα πρέπει να περάσει από το Πάρκιο Άγριας Χλωρίδας και Πανίδας στη Σιέρα Αντεραθένα. Γνωρίζετε ότι πρόκειται για ε, τμήμα του ε, Natura 2000 και είναι πολύ σημαντικό για την ε, βιόσφαιρα. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση δικτύπου, και αυτό που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λόγω του ενδιαφέροντος που έχει αυτό το φυσικό πάρκο θα πρέπει να παραμείνει κατά την άποψή μου ανοιχτή αναφορά και να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα και να λάβουμε και τις πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γνωρίσουμε τι θα γίνει. Ε, το κρατούμε. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Ε, πάλι από την Ισπανία. Ε, σχετικά με, συστάσεις που αφορούν στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διατήρηση του προστατευόμενου από το δίκτυο Natura 2000 πάρκου Λαγκερία στα Κανάρια νησιά. Ε, πάλι η κυρία Δεφάρια παρακαλώ. Yes. Um, the... Ναι, η Επιτροπή ανέφερε ε, ανακοίνωση το Φεβράριο του 2011 σε αυτή την αναφορά και στο μεταξύ πήραμε κάποιες πληροφορίες από τον αναφέροντα και ένα αντίγραφο του χωροταξικού σχεδίου που είχε εγκριθεί για αυτή την περιοχή και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα περισσότερα θέματα έχουν να κάνουν με τη χρήση της γης και όχι με τις αξίες της Natura 2000. Το σχέδιο χρήσης γης αφορά ιδιαίτερα τα θέματα που θίγει ο αναφέρον και σε κάποιο βαθμό επίσης κάποια θέματα διαχείρισης που είναι σημαντικά για τα πτηνά και την χλωρίδα και την πανίδα στην προστατευόμενη περιοχή. Την άλλη πλευρά, το άλλο θέμα που εγείριο αναφέρον έχει να κάνει με τη διαχείριση του χώρου. Εδώ θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η Κομισιόν είχε ανοίξει μια υπόθεση εναντίον της Ισπανίας ε, για τη διαχείριση χώρων Natura 2000 ε, στην περιοχή Μακαρονέζια, διότι σε αυτή την περιοχή η Ισπανία θα έπρεπε ήδη να είχε θέσει σε εφαρμογή μέτρα προστασίας. Γιατί αυτοί οι χώροι έχουν οριστεί ως προστατευόμενοι πριν από έξι χρόνια. Για την ώρα πιστεύουμε ότι το θέματα τα διαχείρισης θα τα παρακολουθήσουμε σε, ε, στην υπόθεση που παραβάσει που χειρίζεται η Κομισιόν. Τα άλλα θέματα έχουν ε, τύχη χειρισμού ε, με το χωροταξικό σχέδιο, το σχέδιο χρήσης γης που έχει ήδη εγκριθεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. χαίρομαι που είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη διαδικασία επί παραβάση, διότι δεν μιλάμε για κάτι τυχείο. Το νησί του Λανθαρότε πλήττεται από μια πολύ σημαντική οικιστική επίθεση, τα δικαστήρια καθυστέρησαν ε, σχέδια για κατασκευή μικροξενοδοχείων και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το φυσικό πάρκο γιατί προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000 και επιπλέον είναι μια ειδική ζώνη προστασίας, ε, χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρά προκειμένου να ε, τηρηθούν όλες οι οδηγίες και θεωρώ ότι και εδώ θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό το ζήτημα για να μπορέσουμε να δούμε και πώς παρακολουθεί το ζήτημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προχωρούμε στην επόμενη, την κρατούμε ανοιχτή, προχωρούμε στην επόμενη, πάλι από την Ισπανία, αναφορά του κυρίου Φραντσέσχο Μέζα Ντιάς, σχετικά με τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στο Εθνικό Πάρκο Ντονιάνα. Και, ε, ναι, και του κυρίου Χαβιέ Καστροβιέιο, ε, ε, εν ονόματι της, της Λέσης της Δονιάνα για τις ε, ε, ε καταστάσεις ερήμωσης στο Εθνικό Πάρκο της περιοχής. από, το, από την Επιτροπή η κυρία Μικελίνη για την πρώτη αναφορά ή ο κύριος Ερνάντες για τις δύο αναφορές. Α, το, το Α, το gracias. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Για την αναφορά αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έκανε ανακοίνωση για την Επιτροπή σας και σας ανέφερε ότι τα περισσότερα από τα θέματα τα οποία καταγγέλλονται έχουν σχέση με αστική ανάπτυξη που δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως γνωρίζετε. Τα περισσότερα από τα θέματα αυτά ούτως ή άλλως είναι αρμοδιότητα των Ισπανικών αρχών. Προσφάτως ο αναφέρον απέστειλε νέα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι στα πρώτα στοιχεία τα οποία μας είχε αποστείλει δεν υπήρχε καμία συγκεκριμένη αναφορά σε ε, παρατυπίες σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στα νέα στοιχεία τα οποία μας έστειλε υπήρχε αναφορά στο πρόγραμμα Ντονιάνα δεύτερη φάση για την περίοδο 94-95 το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΦΕΝΤΕΡ. Επιπλέον, ο αναφέρον μας ε, αποστέλει μία σύνοψη ε, από μία έκθεση του Κοινοβουλίου της Ανδαλουσίας. Δεν έχει ημερομηνία, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για το 2004 και αναφέρεται σε ένα διεθνές κέντρο ε, περιβαλλοντικών μελετών που είναι ένα κέντρο το οποίο κάνει σεμινάρια και συναντήσεις για θέματα περιβάλλοντος στα, στις εγκαταστάσεις του φυσικού πάρκου και ε, μία, και βρίσκεται κοντά στο Δήμο που διαμένει ο αναφέρον. Σε αυτή τη σύνοψη λοιπόν που έχουμε από το Κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας ε, γίνεται μία αναφορά μόνο στις χρηματοδοτούμενες ε, πράξεις και έλεγε απλώς ότι δεν υπάρχει μία αναμνηστική πλακέτα που έλεγε ότι είχε συγχρηματοδοτηθεί το έργο. Πλέον υπάρχει αυτή η αναμνηστική πλακέτα και επομένως το πάρκο λειτουργεί απολύτως και υπάρχουν όλα όσα πρέπει. Ε, το πρόγραμμα τώρα Ντονιάνα ε, για τα όσα έχουν συμβεί για το 94-95 είχε ολοκληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι εκθέσεις ελέγχου, είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι πιθανές παρατυπίες και το πρόγραμμα έχει ε, θεωρηθεί ότι περατώθηκε και όσον αφορά τώρα το ΦΕΝΤΕΡ που είναι το μόνο ταμείο το οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα από τον αναφέροντα, εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και καμία παρατυπία η οποία να μας δίνει ε, το έναυσμα για κάποια περαιτέρω έρευνα επί του θέματος από πλευρά μας. Τώρα θα δώσω το λόγο σε συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας που θα μας μιλήσει με τα γεωργικά θέματα, για τα γεωργικά θέματα της υπόθεσης. Ευχαριστώ. Για το γεωργικό μέρος αναφέρουν, κάνει αναφορά και στο πλάνεμο τεμερίς μας. Ε, συγκεκριμένα παρουσιάζει διάφορα έγγραφα και από κόμματα από τον τύπο που αναφέρονται σε καταγγελίες που έγιναν προηγουμένως από τον κύριο Χουάν Γκαμερατζέα. Ο κύριος Γκαμέρα είναι αντιπρόσωπος ε, κάποιων τοπικών συνεταιρισμών που ε, ισχυρίζονται ότι επηρεάζονται από παραβιάσεις του σχεδίου που φέρονται να έχουν κοινή από τις τοπικές αρχές. Η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει αυτές τις ισχυρισμού και του έχει χειριστεί στο πλαίσιο μιας απάντηση στην ερώτηση 1976 κάθετος 08 και στο πλαίσιο της αναφοράς 0262 του 2008 παρουσιάστηκε από τον κύριο Καμέρο. Η νέα αναφορά που έχουμε τώρα ενώπιον μας δεν ε, γύρει νέα στοιχεία κατά την άποψή μας σε ό,τι αφορά τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά και παρατυπίε. Συνεπώ όπως είπε ο συνάδελφος, διατηρούμε τι παρατηρήσεις που έγιναν ήδη στο παρελθόν, δηλαδή δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι εξ όσων γνωρίζουμε και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, οι ισχυρισμοί που έγιναν σχετικά με το σχέδιο Αλμόντε Μερίς δεν σχετίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια και κατά δεύτερο λόγο η ερώτηση θα πρέπει να τύχει χειρισμού υπό εγχώρια νομοθεσία, εθνική νομοθεσία. Ναι, κυρία Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η Επιτροπή απάντησε και για τι δύο αναφορέ, γιατί νομίζω ότι αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικέ αναφορέ, παρά το γεγονό ότι τι αντιμετωπίζουμε στο ίδιο σημείο, Άλλο είναι το ε, σχέδιο για το Πάρκο Ντονιάνα και άλλο η αναφορά για την επιδείνωση των συνθηκών στο Εθνικό Πάρκο Ντονιάνα. Εσείς αναφερθήκατε αρχικώς στο σχέδιο για το Μόντε Μαρίσμες και καλώς κάνατε, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δεύτερη αναφορά. Ε, ναι, καλημέρα σας. Για τη δεύτερη αναφορά τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την αναφορά έλαβε και αρκετές διαμαρτυρίες από οργανώσεις αλλά και από πολίτες μεμονωμένους, από μία ε, για το Πάρκο Ντονιάνα, καθώς επίσης και μία ερώτηση από τον Βίλι Μέγερ, ο οποίος είναι παρόν εδώ, ε, για τη σχέ, κατάσταση του φυσικού πάρκου Ντονιάνα, το οποίο θεωρείται χώρος ε, κοινοτικής σημασίας, και θεωρείται ότι παραβιάζεται η οδηγία για τους φυσικούς ε, ε, οικοτόπους. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρώτη, ζήτησε πληροφορίες για το θέμα αυτό και τον πιλότο του 2009 στις Ισπανικές Αρχές. Ανατηλήθηκαν οι απαντήσεις των Ισπανικών Αρχών γιατί θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε κατά πόσον θα πρέπει να λάβουμε περαιτέρω πληροφορίες για διάφορες πτυχές, κυρίως όσον αφορά την οδηγία για τους οικοτέσιο για τα ύδατα τις οποίες επικαλούνταν ο αναφέρον και η απάντηση που λάβαμε από τις Ισπανικές Αρχές και αυτή τη στιγμή ε, αναλύεται από τις τεχνικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αλήθεια ότι έχει καθυστερήσει λίγο το θέμα αυτό, αλλά η καθυστέρηση οφείλεται στην πολυπλοκότητα της καταγγελίας, την ε, πληθώρα πληροφοριών που λάβαμε και το γεγονός ότι είναι αρμοδιότητα πολλών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Μέγερ, ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Για τη δεύτερη αυτή αναφορά θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρέμβασή της ε, διότι το φυσικό πάρκο του Ντονιάννα είναι παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO και επομένως η Ευρώπη θα πρέπει να επαγρυπνεί προκειμένου το πάρκο αυτό της Δονιάνα να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή βιόσφαιρα αλλά και για τη διεθνή βιόσφαιρα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό το ερώτημα για τη δεύτερη αναφορά. Ε, <clears throat> δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε με την πρώτη. Να κλείσουμε την πρώτη που αφορά στα funds uh, keep on the second. Και να κρατήσουμε το δεύτερο μέρος ανοιχτό. Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά τα στοιχεία και κοιτάζω τον κύριο Μάιορ τώρα ότι μπορούμε να κλείσουμε την πρώτη αναφορά και να κρατήσουμε ανοιχτή τη δεύτερη. Κλείνουμε την πρώτη και αφήνουμε ανοιχτή τη δεύτερη λοιπόν. Μικρόφωνο παρακαλώ, το μικρόφωνο. με αναφέροντο τον κύριο Ινάκη Ρεγέρο Κάστρο σε ό,τι αφορά τις, ε, σε ό,τι αφορά παραβίαση των οδηγιών για τους οικότοπους και τα άγρια πτηνά ε, στο πάρκο Πίκος de που είναι πάρκο Άγριας Πανίδας, από τις Ισπανικές Αρχές. Ε, η κυρία Έστερ Χορτέτ, από την Επιτροπή. Sí, muchas gracias. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ένα διαδικαστικό ζήτημα. Απαντάμε σε κάποιες συμπληρωματικέ πληροφορίες οι οποίες ε, λήφθησαν τον Οκτώβριο του 2009 για την ε, αναφορά δύο ε, 2006-0166 του κυρίου Ινιάκη Ρεγέρο Κάστρο και όχι για την αρχική αναφορά του 2006 στην οποία είχαμε απαντήσει και είχαμε πει ότι δεν υπήρχε παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που δόθηκαν τον Οκτώβριο του 2009 ε, καταγγέλουν ε, λανθασμένη χρήση κοινοτικών κονδυλίων για το Περιφερειακό Πάρκο του Πίναρ ε, Πίκος Ευρώπα. Και λέγεται ότι δεν Υπάρχει καλή χρήση των κονδυλίων, υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για το πάρκο και ζητά να ληφθούν μέτρα για τις ε, ε, εγκαταστάσεις καθαρισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι το 1994-1995 χρηματοδοτήθηκαν αυτοί οι καταστάσει καθορισμού από το Ταμείο Συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωση. και επίσης θα ήθελαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αναφορά αυτή συμπίπτει με μία καταγγελία που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 με τον ίδιο στόχο και από τον ίδιο αναφέροντα, τον κύριο Ινιάκη Ρεγέρο. Καταρχά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ενημερώσει του. ε, ε ευρωβουλευτές ότι αυτές οι καταστάσεις καθαρισμού είχαν συμπεριληφθεί σε ένα έργο του 1997 και έλαβαν πληροφορίες για να κλείσει το έργο το 2002. Έκλεισε τον Ιούνιο του 2002 και υπήρχε μία έκθεση που έλεγε ότι αυτές οι υποδομές καθαρισμού ε, ήταν πλέον σε λειτουργία. και συνάδουν και με τα όσα πρέπει να ληφθούν βάσει του κανονισμού που προβλέπεται από τον 1164 που αφορά τις ε, διατάξεις του Ταμείου Συνοχής που λέει ότι θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες πριν κλείσει ένα σχέδιο. Από το 2006 ε, που ε, υπευλήθη η αναφορά ε, μέχρι ε, του ΔΕ έχουν γίνει αρκετές επαφές για να δούμε αν αυτές οι υποδομές καθαρισμού ήταν σε λειτουργία. Το πρώτο που μας ελέγχθη ότι ήταν, ήταν ότι ήταν πολύ δαπανηρή η διατήρηση αυτών των υποδομών καθαρισμού. Ε, κατόπιν υπογράφησαν κάποιες συμβάσεις με το Δήμο και, τον, ε, και τους αρμόδιες αρχές του πάρκου για να διαχειριστούν από κοινού διαχει... τα θέματα αυτά. Παρόλα αυτά διαπιστώθηκε ότι οι υποδομές καθαρισμού εξακολουθούσαν να μην λειτουργούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τι ε, Ισπανικέ αρχέ, οι οποίε το Μάιο του 2010 έστειλαν κάποιε τεχνικέ εκθέσει που έλεγαν ότι οι μονάδε αυτέ ε, στην πλειονότητά του λειτουργούσαν μετά από κάποιε εργασίε συντήρησης το 2009. Βάσει τη αρχή τη εταιρική σχέση και τη συνεργασία, μετά από αυτέ τι τεχνικέ πληροφορίε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνθηκε στον αναφέροντα για να κλείσει την αναφορά με τις πληροφορίες αυτές τον Οκτώβριο του 2010. Ο αναφέρον όμως μας είπε ότι πολλές από τις υποδομές καθαρισμού και πάλι δεν λειτουργούσαν. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από τις Ισπανικές Αρχές να κάνουν μια επίσκεψη η οποία θα γίνει τον Ιούνιο για να δούμε αυτές τις υποδομές καθαρισμού και να διαπιστώσουμε επιτόπου κατά πόσον λειτουργούν. Από πλευρά ε, περιφερειακή πολιτική, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι έχει γίνει κάποια παραβίαση, γιατί όταν έκλεισε το σχέδιο, ε, οι μονάδε καθορισμού λειτουργούσαν και δεν υπήρχε καμία παραβίαση. Ε, από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι το κόστος το οποίο δόθηκε το, ε, μας επιτρέπει να κάνουμε έναν επιπλέον έλεγχο επιτόπου για να δούμε κατά πόσον λειτουργούν αυτές οι υποδομίες καθορισμού με συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εσείς στην Επιτροπή σας. Και θα ενημερώσουμε φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από την επίσκεψη στις υποδομές καθαρισμού για να δούμε τι γίνεται με την αναφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μέγερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καθόλου ικανοποιητική. Είμαστε στο σωστό δρόμο, διότι αναφερόμαστε σε μία ε, μοναδική περιοχή της Ισπανίας, το Πίκος Ευρώπα. Και καταρχάς ε, θα ήθελα να πω ότι η αρμόδια αρχή, δηλαδή ο Δήμος της Καστίγια και Λεών ακόμα δεν μας έχει ε, δώσει ε, τι γίνεται με τα σχέδια και διαχείρισης των υποδομών αυτών καθαρισμού και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε ε, ένα μήνυμα από πλευράς Επιτροπής μας ε, που θα διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν έχει ακόμα ε, ανακηρύξει η ζώνη ειδικής προστασίας στο πίκος Ευρώπα ο Δήμος της Καστίγια και Λεόν και δεν έχει λάβει υπόψη ε, πόσο μοναδικό είναι το πάρκο αυτό για τη βιοποικιλότητα της Ισπανίας. Όσον αφορά τώρα τις πληροφορίες που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για η αναφορά κατά την άποψή μας θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, αλλά θα ήθελα να προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα κάνει την επίσκεψή της τον Ιούνιο να μην επαληθεύσει μόνο αν λειτουργούν ε, οι υποδομές καθαρισμού, αλλά επίσης να μεταβεί στους Δήμους ε, της Οθέχα και της ε, Σαχάμπρε, διότι αυτοί οι δύο Δήμοι που βρίσκονται στην, ε, στο πίκος Ευρώπα ε, ρίχνουν τα ε, υδάτινα απόβλητα απευθείας στις εγκαταστάσεις του πάρκου. Θα ήθελα λοιπόν να επισκεφτείτε και το Θέχα Σαχάμπρε για να επιβεβαιώσετε ότι αυτά οι δύο Δήμοι ρίχνουν απόβλητα χωρίς καμία επεξεργασία ε, στο ποταμό ε, στην περιοχή. Λάβει Επιτροπή Μα λείπουν πολλέ πληροφορίε. υπάρχουν ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά για την ώρα μέχρι να εξασφαλίσουμε τις απαντήσεις. Δεν ξέρω αν κατάλαβα σωστά τον κύριο Μάιερ ε, σχετικά με μία δήλωση προς τι αρμόδιες τοπικές αρχές. Νομίζω είναι πολύ νωρί γι' αυτό. Είμαστε ακόμη στα μέσα της διαδικασίας, ε, περιμένουμε απαντήσεις και εδώ στην Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να συζητήσουμε που θα πάμε από εδώ και πέρα. Ας αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να περιμένουμε για τις απαντήσεις. Όταν τις πάρουμε τότε μπορούμε να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Εγώ ήθελα, κύριε Γιάρ, να μου πείτε τι πρόβλημα υπάρχει, γιατί δεν μπορούμε να αποτανθούμε στην περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίγια Ελαιών και να ρωτήσουμε απλώς εάν προβλέπει η περιοχή να ανακηρύξει ζώνη ειδικής προστασίας ε, το Πίκος de Europa. Παρά το γεγονός ότι είναι ισπανική η περιοχή, ε, είναι τμήμα της βιοπικιλότητας όπως η Άλπη, στα Πυρηναία. Επομένως, μία ερώτηση θα μπορούσαμε να κάνουμε. Τι δράσεις σκοπεύουν να αναλάβουν για να προστατεύσουν την περιοχή Πίκος de Europa. Δεν ε, ε, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα και μπορούμε να το κάνουμε στα πλαίσια της παρακολούθησης του θέματος. Ναι, αλλά για το ποιο σύστημα θα εφαρμόσουμε. Χθε αποφασίσαμε να στείλουμε μία σειρά από επιστολές, αλλά πιστεύω ότι είμαστε ακόμη στα ενδιάμεσα της διαδικασίας, όπου δεν έχουν ακόμη απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις μας και τις περιμένουμε ακόμη τις απαντήσεις και είναι θέμα της Επιτροπής. Βέβαια η Κομισιόν το σημειώνει, αλλά στο στάδιο αυτό είναι παρκές να συνεχίσει ο διάλογος ανάμεσα στην Κομισιόν και το κράτος μέλος, αλλά αν έχουμε ερωτήσεις προς τις τοπικές αρχέ θα πρέπει να αποφασίσουμε την άλλη φορά όταν θα πάρουμε τις απαντήσεις. Προσπαθώ να εισαγάγω ένα σύστημα εδώ. Το πρώτο στάδιο είναι να υπάρχει διάλογος ανάμεσα στην Κομισιόν και την Επιτροπή Αναφορών και μόνο όταν εξασφαλιστούν οι απαντήσει, και έχουμε ακόμη ερωτήσεις που θέλουμε να απευθύνουμε τότε να τι στείλουμε στο κράτο μέλο τι θα ήταν η καλύτερη διαδικασία που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Τώρα όμω η Κομισιόν έχει σημειώσει τι αντιρρήσει και τι δικέ σας αντιρρήσει, κύριε Μαΐρ, και μπορούν να επέμβουν αν είναι θέμα της Επιτροπής. Δεν ξέρω αν πρέπει εμεί να στείλουμε επιστολή ε, συνάδελφε ή γιατί Επιτροπή έχει την υποχρέωση να το κάνει αν καταλαβαίνω καλά σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη, τον ορισμό του εν λόγω τόπου ως ειδική ζώνης διατήρησης. Επομένως η Επιτροπή πρέπει να το επιβάλλει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται εμείς να στείλουμε μια συγκεκριμένη επιστολή και να ρωτήσουμε αν έχει γίνει ή όχι. Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη, νομίζω, να το, να το πράξει και να μας ενημερώσει σχετικά. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρά για το βασικό ζήτημα που είναι οι υποδομέ καθαρισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μα είπε τίποτα για το κατά πόσον θα πρέπει να ανακηρύξουμε την περιοχή ζώνη ειδική προστασία, γιατί δεν είναι και αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. το κράτο μέλο είναι αρμόδιο γι' αυτό. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να επισέλθει σε αυτό το θέμα. Θα ασχοληθεί μόνο με τι υποδομέ καθαρισμού. Ποιο είναι αρμόδιο για να διακηρύξει τις, ε, την περιοχή Πίκος ε, Ντε Ευρώπα ε, ζώνη ειδική προστασίας, η Ισπανία. Δεν καταλαβαίνω γιατί διστάζεται. Μπορούμε κάλλιστα να στείλουμε μία επιστολή και να ρωτήσουμε εάν προβλέπουν να ανακηρύξουν ζώνη ειδική προστασία ε, στο πίκο του Ευρώπου. Εάν δεν θέλετε εσεί εγώ ω ευρωβουλευτή, θα στείλω μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ρωτήσω αν θεωρείτε ότι μια περιοχή όπως η Άλπη, τα πυρηνέα ή το Πίκος Ευρώπα πρέπει να θεωρούνται ζώνες ειδικής προστασίας. Και η απάντηση που φαντάζομαι ότι θα μου δώσουν είναι ναι και τότε θα μπορέσω να στείλω μια επιστολή στην ε, Περιφερειακή Κυβέρνηση της Καστίγια Τελεών γι' αυτό. Την πρότασή σας σε ό,τι αφορά τη δική μας ερώτηση, αλλά στο κείμενο που έχω μπροστά μου, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει τις αρμόδιες τοπικές αρχές για το αν έχουν ανακηρύξει ως όφυλαν τον τόπο ως ειδική, ε, ειδική ζώνη διατήρησης. Ούτως ή άλλως η Επιτροπή πρέπει να το κάνει. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι αν παράλληλα με την ε, Επιτροπή που πρέπει να ρωτήσει πρέπει να στείλουμε και εμείς ως, ως Επιτροπή ε, Αναφορών στις ε, ίδιες αρχές μια ερώτηση. Εκεί είναι το ερώτημα το δικό μου. Ε, σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στην Κομισιόν. Ως μέλη ε, βέβαια μπορούμε να θέτουμε ερωτήματα, αλλά η Επιτροπή Αναφορών δεν πρέπει να στείλει μια επίσημη επιστολή στις αρμόδιες αρχές. Είναι θέμα της ε, Κομισιόν, είναι δικό τους καθήκον. Και μετά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όταν εισαλεί. Ε, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής κάποια σχόλια σε αυτά που κουβεντιάζαμε τώρα. Αν δηλαδή είναι μέσα στις υποχρεώσεις της να ρωτήσουν για το αν προκυρεί... Ναι, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ τη Γενική Διευθύνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφού μου δίνεται η ευκαιρία θα ήθελα να το διευκρινίσω το ζήτημα. Η περιοχή Πίκος Δευρώπα, όπως και άλλες περιοχές κοινοτικής σημασίας, βρίσκονται στο δίκτυο Natura 2000. Η οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους, η 2243, καθορίζει μια σταδιακή διαδικασία μέσω της οποίας έξι χρόνια αφότου εγκριθεί ο κατάλογος της βιογραφικής ε, περιοχής που αντιστοιχεί σε αυτή την περίπτωση ε, της βιογραφικής περιοχής του Ατλαντικού, θα πρέπει να καθοριστούν οι αντίστοιχες περιοχές ως ζώνες ειδικής προστασίας. Να δοθεί δηλαδή μια επιπλέον διαβάθμιση ε, στην προστασία που δέχεται η συγκεκριμένη περιοχή. Ο κατάλογος για τις περιοχές του Ατλαντικού εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των ε, ε, Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 2004 και επομένως η προθεσμία εξέπνευσε των 6 ετών το 2010. Άρα το γεγονός ότι η περιοχή Πίκος Δεωρόπα θα είναι ζώνη ειδικής προστασίας είναι ε, εν εξελίξη, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση για την Ισπανία και για κάποιες άλλες χώρες στη διαδικασία αυτή, γιατί το να καθορίσει κάποιος ως ζώνη ειδική προστασίας ένα χώρο δεν είναι μόνο για λόγους σημασίας και ορολογίας, αλλά σημαίνει ότι και το κράτος μέλος θα έχει κάνει και κάποια μέτρα διαχείρισης και ρύθμιση των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να γίνονται στην περιοχή. Στην Ισπανία αυτό γίνεται μέσω των ε, σχεδίων διαχείρισης των φυσικών πόρων και χρήσης και διαχείρισης ε, ενός τοπίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι, γνωρίζει αυτή την καθυστέρηση και θα ήθελε να κάνει όμως μία οριζόντια αντιμετώπιση του θέματος, πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία πληροφόρησης από τα κράτη-μέλη που τους αφορά συγκεκριμένη ε, ανάθεση και αυτή τη στιγμή λάβει τις πληροφορίες εάν ακόμα οι περιοχές δεν έχουν καθοριστεί ως ε, Περιοχέ ζώνες ειδική προστασίας θα ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Επιτρέψτε με να σας πω ότι υπάρχει και προηγούμενο με την πρώτη βιογραφική περιοχή που ήταν ε, η περιοχή Μακαρονέσικα το 2001 που είναι πιο μικρή και πιο περιορισμένη και αφορά μόνο την Ισπανία και την Πορτογαλία διότι μιλάμε για τα ε, σκαναρίου νήσους και τη Μαδέιρα και τι Αζόρες και επειδή η Ισπανία και η Πορτογαλία ε, είχαν καθυστερήσει και πάλι για τη ε, ανακήρυξη των ζωνών ειδική προστασίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία επιπαραβάση λίγο αργότερα κατά των δύο κρατών μελών, διαδικασία επιπαραβάση η οποία εκκρεμεί ακόμα για την Ισπανία και βρίσκεται στο δικαστήριο υπόθεση. Επομένως, η Επιτροπή Αναφορών και οποιοδήποτε Ευρωβουλευτή, εάν θεωρεί ότι απαιτείται, μπορεί να αποτανθεί στο κράτο μέλο, να του υπενθυμίσει την καθυστέρηση και την ανάγκη να τηρήσει το κοινοτικό δίκαιο σε θέματα περιβάλλοντο. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πρέπει να το στείλουμε το γράμμα για να μην ε, ε, ξεχάσουμε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα έτος καθυστέρησης ε, μας δικαιολογεί και μπορούμε με ευγενικό τρόπο να αποστείλουμε επιστολή στις αρχές της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίγελαιών και να τους ρωτήσουμε γιατί έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο. Δεδομένου ότι έλαβα λοιπόν αυτές τις πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ασχολείται εκ παραλλήλου με το θέμα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή μας, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, πρέπει να αποτανθεί στις αρμόδιε αρχές για να μα ενημερώσουν και να μας πούν γιατί έχει καθυστερήσει ένα χρόνο η εφαρμογή τη κοινοτική νομοθεσία. Έχουμε μια πρόταση. Η πρότασή μου, ως συμβιβασμός παρόλο που δεν είναι όλες οι ομάδες ε, παρούσες, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε στην συνεδρία των συντονιστών. Μπορούμε να το κάνουμε ως Επιτροπή, αλλά μετά χρειάζεται η έγκριση όλων των ομάδων και δεν είναι όλες εδώ παρούσες. Ίσως θα πρέπει να συζητηθεί στη συνεδρία των συντονιστών. Αλλιώς να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και η Κομισιόν δουλεύει μαζί μας, χέρι με χέρι, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αναβάλουμε το προφανές. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν η Επιτροπή μας ε, πρέπει να επαγρυπνεί για την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για όλα τα θέματα, αλλά κυρίως για την προστασία φυσικών οικοτόπων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο στην εφαρμογή, και κυρίως για ένα φυσικό οικότοπο, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο και να είμαστε εισάξοι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να στείλουμε μια απλή επιστολή για να ε, ρωτήσουμε όχι μόνο την Ισπανία για, αλλά και άλλους, γιατί όπως μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα κράτη-μέλη έχουν καθυστερήσει για αυτές τις περιοχές οι οποίες είναι ζώνες, θα έπρεπε να ανακηρυχθούν ζώνες ειδικής προστασίας. Γιατί πρέπει να αναβάλουμε την απόφαση για μια απλή επιστολή. Δεν έγινε και τίποτα πια νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε μία επιστολή ευγενική στην ε, Περιφερειακή Κυβέρνηση της Καστίγια Λεών για να μάθουμε γιατί προς τι η καθυστέρηση. Also ich, äh, wenn man sich umguckt, mein Problem ist ein anderes. Ich möchte schon als ε, Πιστεύω ότι εγώ μιλάω για ένα διαφορετικό πρόβλημα. Αν ε, χρειαζόμαστε όλες τις πολιτικές ομάδες ως Επιτροπή να υποστηρίξουμε αυτή την επιστολή και δεν είναι όλες παρούσες. Ε, αυτό έλεγα προηγουμένως και αν το αναβάλουμε δεν θα είναι και καταστροφικό. Ε, γι' αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε στην συνεδρία των συντονιστών όταν όλες οι ομάδες είναι παρούσες. Και ανεξαρτήτως του τι θα κάνουμε, ε, νομίζω έτσι είναι καλύτερη διαδικασία. Αυτή είναι η δική μου σοβαρή απέτηση. Είναι λόγω της προσέλευσης ε, σήμερα το πρωί. Γι' αυτό κάνω αυτή την ε, πρόταση. Πίτερ Γιάρ, δεν καταλαβαίνω τι λες. Ε, νομίζω είμαστε όλοι οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, οι γκουε, δεν μπορούμε να καθόμαστε εδώ κάθε φορά και να μπλοκάρουμε ένα θέμα, διότι δεν είναι μια ομάδα παρούσα. Και ελπίζω να στείλουμε αυτή την επιστολή, το υποστηρίζω και ε, ε, εάν αυτός είναι ο όρος στο μέλλον δεν θα προχωρούμε ποτέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με την Μάργκρα Τάοκεν. όλε οι ομάδε αντιπροσωπεύονται. Μου φαίνεται υπάρχει πλειοψηφία που επιθυμεί να αποστείλει αυτή την επιστολή. Αυτή η Επιτροπή δεν δίστασε ποτέ όταν αισθανόταν ότι έπρεπε να το κάνει. Αυτό που κάνει η Κομισιόν αναπόκειται στην Κομισιόν. Εμεί είμαστε το Κοινοβούλιο και αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ληφθεί δράση, τότε θα ληφθεί δράση. Όλε οι ομάδε εκπροσωπούνται. Νομίζω υπάρχει πλειοψηφία. Ναι, κύριε. Κοιτάξτε, είμαι αρκετά ε, δημοκρατικό και αν η πλειοψηφία το θέλει, τότε θα το κάνω. Μόνο αν υπήρχε περίπτωση να μην θεωρηθεί ότι είναι ε, μέσα ότι είναι νόμιμο να το κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το επόμενο. Μικρόφωνο. Μάουρα Χίλεν, εξ ονόματος της Ένωσης Ασοσιασιών Αμπούζος Ουρμπανίστικος Διαλμαντσόρα κλπ. σχετικά με τον αντίκτυπο της αστικοποίησης στην κοιλάδα της Αλμαντσόρα. Ε, η αναφέρουσα είναι παρούσα. Παρακαλώ να λάβει το λόγο. Η κυρία Χίλεν. Καλημέρα σας. Μπορώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι η περιγραφή της αναφοράς είναι παραπλανητική. Η αναφορά μας ε, είναι εκ μέρους ατόμων που αγόρασαν κατοικίες ε, καλή την πίστη στην κοιλάδα Αλμανζόρα και τελικά ήταν θύματα ε, ενό χάους πολεοδομίας. Το θέμα της κατάχρησης πολεοδομίας στην Ισπανία είναι πολύ γνωστό και ήταν θέμα διαφορετικό διαφόρων εκθέσεων και ψηφισμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο από το 2006 μέχρι το 2009. Και ωστόσο το πρόβλημα υπάρχει και επιδεινώνεται. Θα μπορούσα να σας δώσω πολλές ε, θλιβερές ιστορίες ε, οικονομικών δυσχεριών και εντάσεων που επέβαλε αυτή η κατάσταση σε χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες. Για να σας δώσω την κλίμακα του προβλήματος. Σύμφωνα με μια έκθεση από τον συνήγορο του πολίτη της Ανταλουσίας το 2000, υπολογίζεται ότι υπάρχουν 300.000 παράνομες ε, ιδιοκτησίες στην αυτόνομη κοινότητα της Ανταλουθία και μόνο. Αλλά υπάρχουν 17 αυτόνομες κοινότητες στην Ισπανία θα μπορούσαμε να υπολογίζαμε ένα εκατομμύριο άνθρωπους ε, και ένα συνδυασμέ, μια συνδυασμένη επένδυση δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή έχει και δείξει κατανόηση σε το στο παρελθόν, αλλά συνεχίσει να ισχυρίζεται ότι μπορεί να παρέμβει μόνο εάν το θέμα αφορά την υλοποίηση ευρωπαϊκής νομοθεσία. Πιστεύουμε όμω ότι αυτό αποτελεί όντω θέμα ε, επίθεση ε, και ε, πλήξεις των θεμελιωδών πυλωνών της Ευρωπαϊκής Κοινο... Ε, νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ε, ατόμων. Πολίτες από άλλα κράτη-μέλη έχουν επενδύσει πολλές χιλιάδες αυτές τις ιδιοκτησίες. Οι επενδύσεις τους διακυβεύονται. Αλλά δεν μπορούν να αποεπενδύσουν ή να εγκαταλείψουν τη χώρα πολλώντας τις ιδιοκτησίες τους γιατί τους έχει λεχθεί ότι η ιδιοκτησία τους είναι παράνομη. Η υπόθεση της οικογένειας Πράιορ είναι πολύ γνωστή διεθνώς. Αλλά υπάρχουν πολλές πολλοί κύριοι και κυρίες prior στην Ισπανία, άτομα που επένδυσαν καλή την πίστη, αλλά τώρα κινδυνεύουν να χάσουν την επένδυσή τους χωρίς καμιά ελπίδα για αποζημίωση ή που ζουν χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρισμό ή που αντιμετωπίζουν την απειλή κατεδάφισης ή που πρέπει να πληρώσουν τα χρέη των εργολάβων ή που δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, ιδιοκτησίας ή με συνδυασμό όλων αυτών των προβλημάτων αυτό δεν είναι, δεν είναι καθόλου κίνητρο για άτομα να επενδύσουν στην Ισπανία, όπως έχουν δείξει αυτές οι επενδύσεις. Η συνθήκη προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών πολίτες από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αγοράσει παράνομες ιδιοκτησίες. Πολλές φορές με την βοήθεια ε, κτηματομεσιτών που δεν είναι ρυθμισμένοι ή εργολάβων, developers που δεν εξαναγκάζονται να συμμορφωθούν με ε, τις δικλείδες ασφαλείας ή ε, δικηγόρους στους οποίους στηρίζονται γιατί ε, τους λένε ότι θα τους παρέχουν την ίδια, ε, ε, τις ίδιες υπηρεσίες όπως και στην οικία χώρα τους. Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προστατεύει τους πολίτες από τις διακρίσεις. Αυτό περιλαμβάνει και την άμεση διάκριση. Και εδώ αυτοί οι επενδυτές προέρχονται από χώρες όπου υπάρχουν ρυθμίσεις ε, και ε, επίπεδα ασφαλείας. Αναμένουν αυτά τα πρότυπα να εφαρμάζονται και στην Ισπανία και δυστυχώς ε, σοκάρονται γιατί διαπιστώνουν αυτό δεν ισχύει. Δυστυχώς ε, υπάρχει ίσως και άμεση διάκριση. Και εδώ αναφέρομαι στις ε, αναφορές του Υπουργού του Αρμοδίου για την Πολεοδομία και τη Στέγαση στην Ανταλουσία, που συζητώντας αυτό το πρόβλημα πρόσφατα αναφέρθηκε σε μια ομάδα ανθρώπων που εγκαταστάθηκαν παρανόμως στην επικράτειά μας. Επίσης, βλέπουμε ένα αριθμό παραβιάσεων της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Χάρτα ε, χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζονται κανόνες ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ε, σύνεπως εφαρμόζεται όταν ερμηνεύεται η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ατόμων. Σε αυτό το θέμα βλέπουμε ότι το δικαίωμα αξιοπρέπειας, στέγης και μία παλωτρίωση χωρίς αποζημίωση έχουν τύχει σοβαρής παραβίασης. Έντιμα μέλη, έχουμε ακούσει πολλά λόγια κατανόησης στο θέμα αυτό, αλλά δεν έχουμε δει πολλή δράση. Δεν θέλουμε μόνο την κατανόησή σας, θέλουμε οι νόμοι της Ευρώπης να έχουν μεγαλύτερο νόημα και όχι μόνο λέξεις σε ένα κομμάτι χαρτί. Θέλουμε οι νόμοι της Ευρώπης να επιλύουν ένα πρόβλημα που τουλάχιστον διαταράσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στη χειρότερη περίπτωση καταστρέφει τις ελπίδες και τα όνειρα πολλών ανθρώπων. Θα κλείσω με την παράκληση στην Επιτροπή να ακούσει τις δηλώσεις της Helen Πάιον, της οποίας η κατοικία κατεδαφίστηκε το 2008 και που αυτή τη στιγμή ζει στον καράζ της. Σας ευχαριστώ. Uh, from the Η κυρία Πράιορ. Ευχαριστώ. Τον ε, Ιούνιο του 2002 ο ένας ε, κατασκευαστής ε, πούλησε έξι περιοχές 10.000 τετραγωνικών με άδεια οικοδομήσεως και ε, υπήρχαν τότε 90 σπίτια στην περιοχή. Εμείς ε, διαλέξαμε ένα σχέδιο, πήραμε ένα ε, κτήμα και ξεκινήσαμε την οικοδομή. Στη συνέχεια όμως ο δικηγόρος μας είπε ότι ο κατασκευαστής είχε λάβει όλες τις αναγκαίες άδειε, αλλά το 2003 ολοκληρώθηκε το σπίτι μας και το Μάιο του 2003 μετακινηθήκαμε στην Ισπανία για, σαν μόνιμοι κάτοικοι, είχαμε νερό, ηλεκτρικό και όλα τα αναγκαία χαρτιά. Είχαν ε, ε, πουληθεί και τα υπόλοιπα οικόπεδα και είδαμε ε, να χτίζονται και τα υπόλοιπα σπίτια. Αλλά το 2004 ζητήσαμε να κάνουμε μία διάσταση διάταξη στην πισίνα μας δεν μας είπαν ότι είχαμε πρόβλημα και μετά το 2005 θελήσαμε να αλλάξουμε το γκαράζ και να κάνουμε ένα εργαστήριο και πάλι μας είπαν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Το Μάιο του 2006 μας έδωσαν ένα γράμμα, μας επέδωσαν ένα γράμμα που μας έλεγαν ότι εντός 15 ημερών έπρεπε ε, να έχουμε καταστρέψει το σπίτι και όλα, να έχουμε απομακρύνει όλα τα μπάζα ιδίες εξόδους διότι είχε ανακληθεί η άδειά μας και ε, μόνο η Χούντα Ντε Ανταλουσία και το Δημαρχείο εκπροσωπώντουσαν ε, δεν μας δώσαν καμία πληροφορία πριν η μετά και ο δικηγόρος μας απευθύνθηκε στο συνταγματικό δικαστήριο για να σταματήσει η κατεδάφιση. Η Χούντα όμως της Ανταλουσίας δεν εισάκουσε. Μας έκοψαν το νερό και το ηλεκτρικό και μας έδωσαν δύο ώρες για να αδειάσουμε το σπίτι με ίδια μέσα. Η ε, ε, ε, ε, συνεχίσαμε δικαστικά στη Μαδρίτη και μας είπαν ότι δεν έπρεπε να έχουν μπει στο σπίτι μας και δεν έπρεπε να έχουν καταδαφίσει την οικία μας. Ε, τώρα βλέπετε το βίντεο. Το συνταγματικό δικαστήριο μας δικαίωσε και μας είπαν ότι δεν έπρεπε, ε, ε, δεν μας έδωσαν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούμε στο δικαστήριο που άλλαξε την απόφαση και οι δικαστές είπαν ότι όλες οι ενέργειες μετά από αυτή την περίπτωση ήταν παράνομες και έπρεπε να ξαναχτιστεί το σπίτι μας και να αποζημιωθούμε. Αλλά η Χούντα δεν ε, δέχτηκε την απόφαση του δικαστηρίου και ζήτησε να κατεδαφιστεί και πάλι το σπίτι οπότε συνεχίζεται αυτή η ε, διένεξη ζούμε στο γκαράζ επί 3,5 ε, χρόνια χωρίς νερό και ηλεκτρικό και ο άντρας μου είναι στο νοσοκομείο μας ζήτησαν ε, λοιπόν να ε, ε, υποστούμε εξετάσεις γιατί δεν δέχονται ότι η υγεία μας έχει πληγεί από αυτές τις καταπιέσεις, καταπονήσεις και δεν έχουμε ακόμη καμία εξέλιξη σαφή. Κομισιόν ο κύριος Γαβριλιάδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Είναι ένα θέμα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, ε, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και ατυχώς σύμφωνα με το άρθρο 51.1 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να ε, ε, ε, ευθύνεται κανείς βάσει της αρχής της επικουρικότητας μόνο στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί απλώς να επέμβει στην Ισπανία μόνο σε θέματα εφαρμογής κοινωτικού δικαίου που δεν έχουν διαπιστωθεί αυτή τη στιγμή. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των αναφερόντων. Μπορούν να απευθυνθούν στο Στρασβούργο έργο άπαξ και ε, εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα στην χώρα όπου υπάρχει το πρόβλημα. Κυρία. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η Επιτροπή αυτή έχει λάβει και άλλες αναφορές αυτού του είδους επί 10 χρόνια. Έχει ακούσει πολλούς αναφέροντες επί του θέματος αυτού. Εγώ πέρυσι έθεσα το ίδιο θέμα δύο φορές στον Ισπανό Πρωθυπουργό ο οποίος μας είπε ότι ε, η Ισπανία είναι ένα κράτος δικαίου. Είναι αυτό όμως κράτος δικαίου. Δεν δέχομαι την απόφαση της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κλείσει τα θέματα διότι τώρα πρέπει να δράσουμε και όχι πλέον να ομιλούμε και παρακαλώ την Επιτροπή αυτή να ε, εκδώσει ένα ψήφισμα όπου θα ζητήσει να μπλοκαριστούν οι λογαριασμοί των εμπλεκομένων μέχρι ότου λυθεί το θέμα διαφορετικά θα ζητήσω από τον ε, Βρετανό Πρωθυπουργό ε, να παρακρατήσει <clears throat> τις εισφορές ε, της χώρας μας εις τον κοινοτικό προϋπολογισμό μέχρι ότου βρεθεί λύση. Είμαστε σε μία περίοδο κρίσεως και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέγνωσε σωστά το πρόβλημα και δεν προσέφερε μία γρήγορη λύση. Η κατάσταση αυτή η οποία συνεχίζεται είναι απαράδεκτη και εμείς σαν εκπρόσωποι των πολιτών πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι η μαρτυρία που μόλις ακούσαμε από την ε, ε, δεύτερη αναφέρουσα είναι το πιο συγκινητικό πράγμα που έχω ακούσει εδώ και εγώ προσωπικά θέλω να της εκφράσω όλη μου τη συμπάθεια. Δεν είναι δυνατόν ε, να βλέπει κάποιος να καταστρέφεται το σπίτι σου και οι οικονομίες σου κατά αυτόν τον τρόπο και συγκινήθηκα πολύ από το βίντεο αυτό. Αλλά είναι είναι θέματα γνώριμα, είναι θέματα που έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και εγώ ενοχλούμαι ιδιαίτερος και θυμώνω ιδιαίτερος να μιλάμε για μια Ευρώπη αξιών, για κράτος δικαίου και στη συνέχεια βλέπουμε ότι το κράτος δικαίου καταπατείται κατά αυτόν τον τρόπο από κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε με δεμένα χέρια και μας λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι είναι ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν δεν μπορεί κανείς να τον επικαλεστεί όταν το χρειάζεται. Και εδώ νομίζω ότι εμπλέκεται ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι η Ευρωπαϊκή Συνθήκη των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βασιζόμαστε στην ελεύθερη αγορά, στην ελεύθερη κοινωνία που βασίζεται στο κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου έχει καταπατηθεί στην Ισπανία και φέρονται σαν ληστές, όχι σαν σοβαροί άνθρωποι. Είναι απαράδεκτο ότι μια ελεύθερη αγορά εξαρτάται από το δικαίωμα ιδιοκτησίας και συμβόλαια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, πράγμα το οποίο έχει καταπατηθεί σε αυτή την περίπτωση και δεν πρόκειται μόνο για αυτούς τους αναφέροντες, όπως ξέρουμε είναι πολλές εκατοντάδες Ευρωπαίων πολιτών, Βρετανών πολιτών από χώρες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισπανών πολιτών των οποίων τα δικαιώματα έχουν αγνοηθεί δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν ε, τις υπογεγραμμένες συμβάσεις. Ε, η Ισπανία είναι μια χώρα όπου, όπου έχουν ε, συναυθεί συμφωνίες αυτές παραβλέπονται και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβει. Θα ήθελα προσωπικά να συμφωνήσω με την άποψη της συναδέλφου Ανδρέας. Πρέπει να γίνει κάτι κάτι ουσιαστικό και ε, να παρακρατήσουμε τη χρηματοδότηση της Ευρώπης από αυτές τις περιοχές. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό, θα το στηρίξω και ελπίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας συνδράμει του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω εμπλακεί με το θέμα αυτό από το 2004 θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μάουρα για την παρουσίασή της και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αναφέρουσες για την παρουσία τους εδώ εν γέννη. Να πω ότι δεν ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και μία δεκαετία, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και οκτώ χρόνια. Η θέση του Κοινοβουλίου υπήρξε σαφής για το τι συμβαίνει από πλευρά τη οργάνωσης, τι γίνεται με την ε, νόμιμη αγορά παράνομων ε, οικημάτων. Ε, είναι απαράδεκτο. Και θα ήθελα να πω στην κυρία Αντρέασον και στον κύριο Χέλμεν ότι οι πτυχέ του προπολογισμού έχουν ήδη ψηφισμοί ψηφιστεί στο ψήφισμα του 2009. Υπάρχουν λοιπόν και γιατί να κάνουμε έκκληση για κάτι το οποίο ήδη υπάρχει. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο. Η χάρτα ισχύει μόνο σε άμεση σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα πρέπει να πω ότι ότι εάν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, αν υπήρχε ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ιδιοκτησίες και την απόδοση δικαιοσύνης για τα θέματα αυτά, θα είχε ε, αποδοθεί δικαιοσύνη το 2004. Δεν σας μιλώ ε, έτσι τυχαία. Επισκέφθηκα εξ ονόματος του Κοινοβουλίου σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις ε, επιτόπου την περιοχή και πραγματικά η προσωπική τραγωδία των ανθρώπων αυτών υπάρχει και υπάρχει για ανθρώπους από όλη την Ευρωπαϊκή ε, όταν λένε κάποιοι ότι είναι βρετανικό το ζήτημα, λανθάνουν. Πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα, διότι υπάρχει το βασικό δικαίωμα, τη ελευθερία μετακίνηση και το δικαίωμα κάποιο να διαμένει και να συνταξιοδοτηθεί και να φυτά και να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Και αυτό λοιπόν είναι ευρωπαϊκό ζήτημα τι πρόβλημα υπάρχει. Από κάποιε πλευρέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο. Μπορούμε να καταφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την οποία θα πρέπει να προσυπογράφει κάθε κράτο μέλο πριν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, η αναφορά αυτή θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, διότι οι δράσει και οι τρέχουσε αλλά και οι προηγούμενε τη Ισπανική κυβέρνηση δεν συμμορφούνται με την Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σαφώς υπάρχει και ε, έλλειψη πρόσβασης ε, σε, στη δικαιοσύνη για αποζημιώσεις. Αυτό είναι αληθές. Επίσης, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, είτε λόγω σχεδιασμό είτε παραδρομή, οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ δεν έκαναν το καθήκον του. Δεν μιλάμε για ε, ε, μία μικρή περιοχή, μιλάμε για έξι σχέδια που το καθένα από αυτά ήταν 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Αν δεν ξέρει τι κατασκευάζεται στην περιοχή σου, τότε δεν προστατεύει το βασικό καθήκον των, ε, που έχει προ του πολίτε σου, που είναι να φροντίζεις το περιβάλλον και όλη την περιοχή για την οποία υποτίθεται ότι ψηφίστηκες ε, να την αντιπροσωπεύεις. Και εδώ ε, θα πρέπει να ληφθούν πολλά μέτρα, να υπάρχει και ένα ε, δικαστήριο για... και αυτό προσπαθώ να καταφέρω με την Ισπανική κυβέρνηση για να μπορέσουμε και με τους υπουργού και με τους περιφερειακούς υπουργού, γιατί το όλο θέμα της περιφερειακής αυτονομίας περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα στην Ισπανία και εμείς από πλευρά Κοινοβουλίου θα πρέπει να ζητήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε είτε με, μια, ε, με ένα αίτημα προς την Ολομέλεια, αλλά... Ε, εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε διαμέσου της Ολομέλειας, θα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τους περιφερειακούς υπουργού και τους εθνικούς υπουργού να συναντηθούν και να παρουσιάσουν, να συστήσουν, συγγνώμη, μία επιτροπή για να δούμε κατά πόσον μπορεί να δοθεί κατάλληλη αποζημίωση για ανθρώπους που αγόρασαν νομίμως, και το νομίμως το τονίζω, της ιδιοκτησία τους μέσω του Ισπανικού δικαστικού συστήματος χρησιμοποιώντας το χωροταξικό σύστημα της Ισπανίας και επομένω, εφόσον έκαναν αγορά εκεί έχουν δικαίωμα και έχουν ένομο δικαίωμα να διαμένουν στην περιοχή. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη άγουσα και θα πρέπει να είμαι ειλικρινής εδώ Είμαστε κοντά σε εκλογές στην Ισπανία. Θα υπάρξουν πολλές υποσχέσεις, θα σας τάξουν πολλά, αλλά πρέπει να σας πω ότι εάν υπάρξει συμφωνία για ε, τη σύσταση της Επιτροπής αυτής από τους Ισπανούς συναδέλφους ε, και τους εθνικούς βουλευτές ε, πριν φτάσουμε στην προεκλογική περίοδο. Εγώ θα το κυνηγήσω προσωπικά, το κάνω με τους Ισπανούς σοσιαλιστές συναδέλφους ήδη ε, μου είπαν ότι η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας εξετάζει το όλο ζήτημα και ε, θέλει να δώσει κάποιο νόμιμα δικαίωμα στις ε, αφαίρετες αυτές κατοικίες. Αλλά αυτό που θέλουμε να είμαστε βέβαιοι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο είναι να πιέσουμε ώστε όλες αυτές οι υποσχέσεις που δόθηκαν σε χαλεπούς καιρούς θα υλοποιηθούν και θα υπάρξει δράση μετά από, την προεκλογική, μετά από τις εκλογές. Συγγνώμη. Και τέλος, να σας πω ότι χαιρετίζω το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ασχολούνται με το ζήτημα. Κάποια πολιτικές ομάδες δεν πιστεύουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να επιληθεί αυτό είναι διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμέσου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την επόμενη φορά που θα δω τον κύριο Μπαρόζο θα το ρωτήσω προσωπικώς τι μπορεί να κάνει ε, τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι επίτροποι πέραν των νομικών του αρμοδιοτήτων για να πιέσουν την Ισπανία. Διότι θα πρέπει να θυμάστε ότι αυτοί που ζητούν δράση θα είναι και οι πρώτοι που θα καταγγείλουν και αναφέρομαι στην ε, ε, κυβέρνηση και στους πολιτικούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ε, σε τομείς που άλλοι θεωρούν ότι δεν έχει νομική αρμοδιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση, να μην υπάρχει πολιτικό ε, όφελος και να μην ε, ασχοληθεί με το πολιτικό ζήτημα κανένας άλλος εκτός από, από τους αναφέροντες. Και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αναφέροντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάσμαν. Η κυρία Άουκε. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και φυσικά ευχαριστούμε την αναφέρουσα που ήρθε εδώ και μας περιέγραψε και λυπάμαι να πω για ακόμη μια φορά δεν θα έλεγα ότι είναι πιο συγκινητική αναφορά γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές ε, στο ίδιο επίπεδο ε, που δεν βελτιώνει τα πράγματα για αυτή την υπόθεση ε, υποστηρίζω πλήρως αυτά που είπε ο Κάσμαν θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημεία πρώτον προς την Κομισιόν Βέβαια, η απάντηση είναι δεν είμαστε εμείς, να προσφύγετε ε, στο ΕΔΑΔ, στο Στρασβούργο και ξέρετε όπως και εγώ ότι αυτή είναι, δεν, ε, είναι, δεν είναι καλή στατική. Παίρνει δεκαετίες στο Στρασβούργο ε, να επιληφθεί μια υπόθεση. Είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα χρόνια χρειάζονται. Θα ήθελα να επενθυμίσω την Κομισιόν ότι μια μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο υπερψήφισαν την έκθεσή μου, που σημαίνει ότι εμείς το Κοινοβούλιο ε, πιστεύουμε ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα και θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα και η Κομισιόν θα πρέπει να σεβαστεί το γεγονός ότι ακόμη και αν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τη χάρτα, ε, όλοι έχουμε ε, μελετήσει τις παραγράφους και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ε, χάρτα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, στη Νέα Συνθήκη, στο άρθρο 2, αναφέρονται βασικές αξίες και αν αυτές οι αξίες δεν είναι αξιόπιστες σε κάποιο βαθμό τότε θα πρέπει να διαλύσουμε αυτό το σώμα τι, τι, αξία έχει αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ε, αξίες ε, που αναφέρονται στην αρχή της συνθήκης. Σας πενθυμίζω, συνάδελφοι, ότι αποφασίσαμε να έχουμε μια ακρόαση για θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων και πώς τα χειριζόμαστε. Διότι είναι πολύ ανιαρό να ακούμε αυτή την απάντηση από την Κομισιόν δεν ε, εναποκείται σε εμά. Δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι. Ναι, είναι και εσεί και εμεί και πρέπει να βρούμε, ίσως να βρεθούν άλλοι νέοι τρόποι και θα πρέπει να πάρουμε κάποια συστάσεις από την έκθεσή μου, όπως ε, αναφέρθηκε και από τον Κάσμαν. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια σημεία. Μπορεί να θυμάστε τι έγινε τον φθινόπωρο του 2009, μετά τις εκλογές. Ε, στο προπολογισμό. μα είχαν ξεγελάσει διότι είχαμε μια σαφή τροπολογία σύμφωνα με αυτά που είχαμε αποφασίσει την εκθεσή μου ότι ε, ιδιαίτερα για την Βαλένσια αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα ε, μέρη. Αν δεν έχουμε σαφείς βελτιώσεις, θα πρέπει να παρακρατείται η χρηματοδότηση μέχρι να δούμε βελτιώσεις. Αυτή η τροπολογία, όμως, εκεί μας ξεγέλασαν και εκεί τέθηκε όχι ένα συμβιβασμό, αλλά ήταν σχεδόν διαδικαστική απάτη αυτό που έγινε για τη δουλειά μας. Θα πρέπει να το ξαναπροσπαθήσουμε, να είμαστε έτοιμοι να ε, επιμείνουμε σε αυτό το θέμα στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών, γιατί ξέρω τι έγινε, ξέρω ποιοι είναι οι πέτοι και υποστηρίζω ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε τα θέματα. Τα... Ε, θα μπορούσαμε επίσης, η Επιτροπή θα μπορούσε να θέσει μια τροπολογία στον προπολογισμό. Στην, ε, στο θέμα του διαμεσολαβητή, του συνήγορου του πολίτη. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ε, καλύτερα. Αλλά αν εμεί ω Επιτροπή ζητήσουμε για μια τροπολογία στον προπολογισμό. Θα δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε αυτό. Δεν είμαι ειδική, αλλά νομίζω είναι δυνατόν. Για να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη δύναμη, διότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Και είναι δεκ, δεκάδες χιλιάδες οι αναφέροντε και η πλειοψηφία είναι ισπανικής ηθαγένειας. Ε, δεν αφορά μόνο τουρίστες και ξένους. Οι περισσότεροι αναφέροντες, τουλάχιστον στη δική μου έκθεση, ήταν Ισπανοί. Να, επίσης και το θέμα ε, του νόμου ε, για τις παρακτίες περιοχές. Υπάρχει ένα ε, σημείο κοινό ανάμεσα σε αυτά τα δύο να ζητήσουμε από το Ισπανικό σύστημα να απαντήσει φέτος. Εγώ το έκανα όταν ήμουν εκεί και σε πολλές υποθέσεις ήταν εμφανές. Γιατί να μην προσφύγουν στα δικαστήρια. Και ο κόσμος είχε θυμώσει μαζί μου. Καταλαβαίνω γιατί. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα να πάει κανείς στα δικαστήρια εκεί. Τα δικαστήρια δεν μπορούν να το χειριστούν, έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας. Και το κόστος επίσης είναι δυσβάσταχτο. Όταν κερδίσεις μια υπόθεση, η ε, ε, ε, άλλη πλευρά είναι ισχυρότερη, μπορεί να το υποβάλει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και τελικά είναι δυσβάσταχτη η κατάσταση. Γι' αυτό θα πρέπει να το χειριστούμε εδώ αυτό το θέμα και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που είναι να ασχολούμαστε με τα βασικά δικαιώματα των ανθρώπων και αυτό είναι δικαίωμα ιδιοκτησίας. Είναι βασικό δικαίωμα. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση ή αναφέρουσα. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ, ευχαριστώ για τους ε, αναφέροντες που μας παρουσίασαν το θέμα αυτό και ε, θα ήθελα να πω να ε, πω εις ε, τους αναφέροντας ότι πάλι καλά που επεβίωσαν από αυτή τη δοκιμασία διότι ε, είδαν το έργο ζωής τους να καταστρέφεται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου είναι πολιτικό. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και δεν έχουμε πραγματικά καμία δυνατότητα να επέμβουμε. Οπότε τότε πολύ σωστά πρέπει να ερωτούμαστε γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν είναι μία επινόηση ανευνοήματος, πρέπει να μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι μία ένωση αξιών και στην περίπτωση αυτή πρέπει να δούμε τι μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε. Ξεκινώ λοιπόν από την προϋπόθεση ότι η Ένωση δεν πρέπει να εξασφαλίσει μόνο ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και των εργαζομένων, να έχουμε κοινέ αξίες για το περιβάλλον, αλλά να διασφαλίζουμε από κοινού και τα δικαιώματα των πολιτών. Και το ελάχιστο κατά τη γνώμη μου είναι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας ιδιοκτησίας και της ελεύθερης διακίνησης αυτής της ιδιοκτησίας. Για μένα αυτό είναι η επικεφαλίδα πάνω από όλε τι αρχές. Στην Γερμανία παραδείγματος χάρη ο ε, ε, πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θεωρώ ότι πρέπει να έχει εμπιστοσύνη όπου κατοικεί, να γνωρίζει ότι προστατεύεται όπου και να είναι η ιδιοκτησία του και το έχω πει επανειλημμένος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κράτος ε, για ε, ε, δικούς τους λόγους πρέπει να ε, επέμβει σε μια ιδιοκτησία αλλά τότε αυτό πρέπει να γίνεται έναντι αποζημιώσεως και η αποζημίωση αυτή είναι και αποτρεπτικό στοιχείο για το κράτος να μην μπορεί να επεμβαίνει στις ιδιοκτησίες χωρίς καμία αποζημίωση είναι παράνομο και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι τι όμως μπορούμε να κάνουμε καταρχήν να μείνει ανοιχτή η ε, αναφορά διότι όταν υπάρχουν σοβαρές ε, παραβιάσεις του δικαιώματος ιδιοκτησίας από τις αναφορές θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτές να γίνει μια σημαντική ακρόαση σε συνδυασμό με τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας έχει πει η νομική μας ε, υπηρεσία ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση αλλά ε, τα θέματα αυτά ε, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και να συμπεριληφθούν στην ακρόαση αυτή την εκτενή την οποία εγώ ε, επιθυμώ και πολιτικά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Εξού και η πρότασή μου. Μέχρι σε αυτού του σημείου συμφωνούμε φαντάζομαι όλοι. Αλλά αυτό που θα πω από εδώ και μπρο είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε και να συζητήσουμε από κοινού ίσως επίπεδο συντονιστών. Δηλαδή, μήπως ε, δεν θα έπρεπε απλώς να προσφέρουμε ελπίδες στους αναφέροντες αλλά να προσπαθήσουμε να λύσουμε και το πρόβλημά τους. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι καταρχήν πρέπει να απευθύνουμε μία πολύ αυστηρή επιστολή σε όλα τα κράτη-μέλη γιατί είναι θέμα των κρατών μελών τα οποία δεν μπορούν ε, να διαφορούν για τα τεκτενόμενα. Ε, δεν φτάνει απλώς να κάθονται με δεμένα χέρια. και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και ε, να συζητήσουμε και με τις ε, ε, άλλες επιτροπές, με τους συναδέλφους οι οποίοι είναι σε παρεμφερείς επιτροπές και πρέπει να δούμε τι γίνεται όταν υπάρχουν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και τι γίνεται από πλευράς δημοσιονομικής. Οι υπόλοιπες όμως παρατηρήσεις μου θα περιοριστούν σε μία συνεδρίαση των συντονιστών διότι κατά τη γνώμη μου πρόκειται για το δικαίωμα ιδιοκτησίας του πολίτη σε κάθε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν με ενδιαφέρει πού υπάρχει το παράπτωμα, μπορεί να είναι γιατί στην Ιρλανδία, μπορεί να υπάρχουν σε άλλες χώρες περιοχές οι οποίες είχαν πλημμυρίσει, πρέπει όμως να μπορεί κανείς να βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προστατεύεται και ε, γίνεται σεβαστό το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και αυτό πρέπει να ισχύσει και σε αυτή την περίπτωση. Ναι, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήθελα καταρχάς να επαναλάβω στις αναφέρουσες ότι συμμερίζομαι το πρόβλημά τους, να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Το είδα και ιδίω όμαση σε μία επίσκεψη επιτόπου και μετά από τη συζήτηση που έκανα με τους αναφέροντες έκανα και ερώτηση νομίζω το 2010 τον Ιανουάριο με, προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι σαφή. Λόγω προβλήματος διαχείρισης και διοίκησης οι πολίτες είναι θύματα κακοδιαχείρισης. Στην περίπτωση της Ισπανίας μιλάμε για ένα θέμα το οποίο άπτεται 30 δήμων. Πολλοί πολίτες, καλή την πίστη, είτε Ισπανοί είτε Ευρωπαίοι πολίτες, έλαβαν άδεια από την ε, τοπική διοίκηση για την κατασκευή κατοικίας, ελάμβαναν την άδεια δόμησης, ε, επομένως αυτοί είχαν τηρήσει τις απαιτήσει, αλλά επειδή οι χωροταξικές αρχές στην Ισπανία είναι ε, και αρμοδιότητα των τοπικών αρχών και των περιφερειακών αρχών, λόγω προβλήματο συντονισμού μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών, είναι θύματα. Γιατί οι πολίτε ε, δεν έχουν κάνει κάτι παράνομο. Όταν ζητούν άδεια και του δίνεται η άδεια θεωρούν ότι τοπική αυτοδιοίκηση ή περιφερειακή διοίκηση τους δίνει όλα τα εχέγια για να κατασκευάσουν την κατοικία τους. Έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή αυτή ε, πάνω από αρκετές χιλιάδες ε, κατοικίες ε, στις περιοχές αυτές. Το σφάλμα δεν είναι των πολιτών αλλά των αρχών που έδωσαν άδειες. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι μία απόπειρα να νομιμοποιήσουν κάποιο ε, ε, αριθμό εξ αυτών των ε, κατοικιών και να καταδαφίσουν 270 αν δεν κάνω λάθος, αν έχω σαφή στοιχεία. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πλήττονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι αναφέρουσες έγιναν θύμα, θύματα εν μία νυχτή και ξαφνικά βρέθηκαν άστεγες λόγω διοικητικού λάθους. Και θεωρώ ότι αυτό είναι απαράδεκτο. απαράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν εμείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ένας πολίτης από οποιαδήποτε χώρα και αν κατέγεται και ε, σε όποια χώρα και αν διαμένει όταν λαμβάνει άδεια από μία αρμόδια αρχή ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει και όλα τα νομικά εχέγγυα ώστε αυτός ο άνθρωπος να μην ε, ε, βρεθεί ένα δίκο και λόγω λάθους της διοίκησης. Συμφωνώ με όλες τις πρωτοβουλίες που προτείνονται και έχουμε και ε, θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει ο καθένας μας δικαίωμα στην κατοικία, καθένας μας ε, δικαίωμα να ε, ε, ξεκουραστεί γιατί το αξίζει όταν ειδικά δίνει όλες του τις οικονομίες για να αγοράσει μια κατοικία η οποία υποτίθεται ότι έχει κατασκευαστεί νομίμως και θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και σε αυτή την ακρόαση που θα κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα να θέσουμε και το συγκεκριμένο ερώτημα ε, για να παρουσιάσουμε και να έχουμε μια βάση από πλευρά μας που να μην επιτρέπει λόγω λάθος των αρμοδίων αρχών να γίνονται θύματα οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουσουτήλ παρακαλώ τους επόμενους ομιλητές να είναι λίγο έτσι φιδωλοί με το χρόνο, ο οποίος τρέχει πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βέβαια έχω συγκινηθεί και εγώ όπως και οι προλαλήσαντες από τα λόγια των αναφέρουσων και θα ήθελα να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου την αλληλεγγύη μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε ότι αν η Κομισιόν πιστεύει ότι δεν υπάρχει παραβίαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε δεν υπάρχει διορθωτικό μέτρο το οποίο μπορούμε να πετύχουμε. Ο πρόσωπο τη Κομισιόν στην απάντηση ήταν πολύ συγκεκριμένο. Αναφέρθηκε στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αναφέρθηκε στο κεφάλαιο ε, συγκεκριμένα κεφάλαιο που να αποδεικνύει ότι δεν είναι εφαρμόσιμο. Αλλά δεν αναφέρθηκε στο θέμα τη ελεύθερη κινήση κεφαλαίων, που ήταν ένα θέμα το οποίο έθιξε η αναφέρουσα. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, εάν θέλω να αγοράσω μια ιδιοκτησία στην Ισπανία και μου λένε ότι δεν μπορώ να την αγοράσω, τότε αυτό αποτελεί παραβίαση τη ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ωστόσο όμω, εάν αγοράσω αυτό το σπίτι και μου το κατεδαφίσουν οι αρχέ, δεν υπάρχει καταβίαση τη ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Θα ήθελα τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν να εξετάσει αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει παραβίαση τη αρχή ελεύθερη διακίνηση. Διότι εάν το, κατεδαφίζεται το σπίτι, μπορεί να μην αποτελεί παραβίαση ε, για εκείνον τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη της κατοικίας αλλά σίγουρα αποτελεί ε, αντικίνητρο για όλους τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες για να αγοράσουν ιδιοκτησία στην Ισπανία. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελούσε ε, παραβίαση. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν αν αυτό το θέμα έχει παραπεμφθεί στο, ε, στο, στο, μάλλον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και αν έχει αποφασιστεί στο δικαστήριο. Αν όχι, δεν θα έπρεπε η Κομισιόν να το παραπέμψει στο δικαστήριο, δεδομένου ότι υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στο θέμα της ερμηνείας του, εάν υπάρχει, αν δεν υπάρχει ε, παραβίαση της διακίνησης κεφαλαίων. Θα ήθελα η Κομισιόν να απαντήσει σε αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τις αναφέρουσες και να, μου ε, είπα να μην ε, εκφράσω τη συμπόνια μου, αλλά θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι αρκετοί σε αυτή την Επιτροπή δούλεψαν πολύ σκληρά στα θέματα αυτά, ιδιαίτερα η κυρία Όκεν και ο κύριος Κάσμαν. Θα ήθελα να του ευχαριστήσω για τη δουλειά που έκαναν, γιατί το παρακολουθούσα, παρακολουθούσα τη δουλειά τους και τους υποστήριζα, αλλά πολλή δουλειά είχε επιτελεστεί. Το θέμα είναι που, προς που θα πάμε από εδώ και μπρος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την Επιτροπή να είμαστε ειλικρινεί με του πολίτες. Να μην φεύγουν από εδώ και να περιμένουν διορθωτικά μέτρα που εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να τους δοθούν. Και έχουμε ακούσει λόγια για δικαιώματα ιδιοκτησία που δεν βρίσκονται στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν βρίσκονται. Και πολλοί αυτοί που λένε ότι θα πρέπει να βρίσκονται αυτά τα δικαιώματα, δεν θα το υποστήριζαν ε, πρώτα-πρώτα. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί σε αυτά που λέμε στου πολίτε. Το θέμα είναι πώ θα προχωρήσουμε από εδώ και μπρο. Κάποιε εισηγήσει έχουν προταθεί. Ίσως ο τελευταίο ομιλητής μίλησε για τη διακίνηση κεφαλαίων. Ίσως να υπάρχουν κάποιε λύσει εκεί. Επίση και η κυρία Όκεν μα είπε για την τροπολογία στο προπολογισμό από πλευράς αυτής της Επιτροπής θα μπορούσαμε εδώ να προχωρούσαμε κάπως. Θα εισηγόμουν να υποστηρίξουμε αυτό. Αλλά πέραν της υποστήριξης θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι θα διασφαλίσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ότι οι ομάδε μας επίσης θα το υποστηρίξουν για να βεβαιωθούμε ότι θα περάσει τελικά. Ο κύριο Κάσουμαν μίλησε για ένα δικαστήριο που ίσως να υπάρχουν ευκαιρίες επίλυσης. Θα δούμε πώς θα γίνει. Εγώ έχω μια τελευταία εισήγηση ε, από μια υπόθεση που είχαμε στην Ιρλανδία για άδεια οικοδομής, πολεοδομίας ε, και η Επιτροπή αποφάσισε αυτό. Σε αυτή τη ρήτρα υπάρχουν περιορισμοί ε, στο άτομο, δηλαδή η άδεια πολιοδομία δόθηκε να οικοδομηθεί μια κατοικία όπου το άτομο έπρεπε να παραμείνει στο σπίτι για μια περίοδο 5 έως 6 ετών. Η Επιτροπή ε, αποφάσισε και είπε στις Ιρλανδικές αρχές και το αμφισβήτησε αυτό. Η βάση ήταν η ελευθερία εγκατάστασης, όχι διανομονής ιδιοκτησίας, αλλά εγκατάστασης, με άλλα λόγια. Εάν ένα άτομο, για παράδειγμα, ήθελε να έχει μια επιχείρηση από το σπίτι, δεν ήταν μόνο για οικιστικού ε, Σκοπούς. Αν ήθελε κάποιο να έχει την επιχείρηση του από το σπίτι, τότε υπήρχε ε, διαφορά εκεί. Και η Κομισιόν ζήτησε από όλε τι τοπικέ αρχέ τη Ιρλανδία να αλλάξουν την νομοθεσία σε αυτό το θέμα. Και περισσότερε στη συνέχεια το έκαναν. Δεν ξέρω αν υπάρχει διασύνδεση εδώ, αλλά λέω ίσω να είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε. Είναι κάτι το οποίο σκέφτηκα από μια προηγούμενη αναφορά. Το αφήνω εδώ και ε, θα δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε από την Κομισιόν στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου φαίνεται ότι τα αυτιά των ε, αρμοδίων αρχών στην ε, Ισπανία θα πρέπει να κοκκινίζουν από ντροπή με αυτή τη συζήτηση. Ντροπή που επιτράπηκε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για τόσο καιρό. Μου φαίνεται ότι αυτή είναι συμπεριφορά όχι μόνο τόσο δημοκρατίας και κράτους δικαίου, αλλά ε, ενός αυταρχικού κράτους, ολοκληρωτικού κράτους και είναι εκπληκτικό να συμβαίνει αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια κατάσταση που είναι πολύ απογοητευτική, έντονα απογοητευτική και ματαιωτική. Ε, έχουμε ακούσει από, από τους συναδέλφους και τι να πούμε για τις αναφέρουσες. Ε, και βέβαια είναι απογοητευτικό διότι φαίνεται να μην μπορούμε να κάνουμε, προχωρήσουμε, να κάνουμε πρόοδο στην επίλυση. Υποστηρίζω φυσικά την πρόταση της κυρίας Άουκεν. Έχει δουλέψει εξαιρετικά σκληρά στο θέμα αυτό και ως Επιτροπή θα πρέπει να κάνουμε μια αποφασιστική προσπάθεια εάν υπάρχει φυσική δικαιοσύνη που θα πρέπει να ε, αποκατασταθεί θα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Ε, έχω σκεφτεί ότι η Ισπανία έχει ένα μεγάλο αριθμό αδειών ιδιοκτησιών ως αποτέλεσμα της ε, πτώσης των ιδιοκτησιών και το ερώτημα είναι γιατί κατεδαφίζουν σπίτια στα οποία ζουν οι άνθρωποι μέσα και αφήνουν άδεια σπίτια ε, Είναι πολύ περίεργη αυτή η λογική και η τελευταία μου ε, σκέψη σήμερα είναι ε, όπως έχουν τα πράγματα ε, δεν με πλήττει το γεγονός ότι άνθρωποι, μια πλειοψηφία των ανθρώπων του Γιβραλτάρ που εκπροσωπώ σε αυτό το κοινοβούλιο δεν έχουν καμιά επιθυμία να έχουν τίποτα να κάνουν με τις, ε, ε, τις αυτό που επιθυμεί η Ισπανία εδαφικά στο Γιβραλτάρ. Οι, Ισπανοί θα πρέπει όμως να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Θα πρέπει να τακτοποιήσουν ε, τις υποθέσεις εντός της χώρας τους και να αποκαταστήσουν την τιμή τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω στο θέμα της εκθέσεως της κυρίας Άουκεν, η οποία λέει ότι μπορεί κανείς να παρακρατήσει κονδύλια εάν δεν έχει λυθεί το θέμα. Και εφόσον δεν έχει λυθεί το θέμα, νομίζω ότι τώρα πρέπει να ενεργήσουμε και να ζητήσουμε να μπλοκαριστούν τα κονδύλια. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια σωστή ενέργεια. Επίσης πιστεύω ότι η κυρία Άουκεν στην έκθεσή της η οποία είχε υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια αλλά δεν υπήρξε μία ομόφωνη απόφαση ακόμη και οι περισσότεροι Ισπανοί βουλευτές είτε ε, απήχαν είτε ε, καταψήφισαν και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κάσμαν διότι Υπάρχουν πολλοί Ισπανοί οι οποίοι πλήττονται με τον ίδιο τρόπο και ε, ε, ε, δεν θέλουν να ψηφίσουν μία έκθεση σαν της κυρίας Σάουκεν. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να είναι δυνατόν να δεχθούν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ πολιτικό και είναι θέμα ευρωπαϊκής συνοχής διότι δεν υπάρχει αξιοπιστία μεταξύ των λαών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ο κύριος Μπουσουτήλ έκανε μία ερώτηση στην ε, Κομισιόν. Είσαστε έτοιμοι να απαντήσετε τώρα. Κύριε Κάσμερ πρώτα όμως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό σας έδωσα την έκθεση Άουκεν, γιατί ε, πρέπει να γνωρίζουμε τι ζητά η έκθεση Άουκεν. Ζητά να καταρτιστεί αυτή η Επιτροπή. Ζητά να αναγνωρίσουμε ε, το Δικαστήριο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, η στο Στρασβούργο και υπάρχει μια Βρετανική εταιρεία η οποία ετοιμάζει μια τέτοια σειρά προσφυγών. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα θέματα που στην έκθεση αυτή που αναφέρεται εις ε, τα δημοσιονομικά θέματα στην ε, παράνομη διάταξη η οποία ζητά να υπάρξει αποζημίωση για τους καταναλωτές οι οποίοι είναι θύματα τέτοιων μεθόδων και ακόμη και αν δεν μπορείτε να αντιδράσετε άμεσα βλέπετε ότι πρέπει κανείς να εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι υπάρχουν κινήσεις που μπορούν να αναλυφθούν μέσω του δικαστηρίου των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ας εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι η έκθεση Άουκεν θα εφαρμοστεί εφόσον έχει υπερψηφιστεί. όσον αφορά την ε, ελευθερία εγκατάστασης. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Προς ποιον θέλετε να κάνετε την ερώτησή σας. Ναι, ναι, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Πιστεύω καταρχήν ότι ο κύριος Κάσμαν πολύ σωστά ε, θύμισε διάφορες αρχές δικαίου οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην υπόθεση αυτή. Μία πολύ βασική αρχή είναι σωστή απροζημίωση για κάποιον ο οποίος στερείται από ένα κράτος μέλος της περιουσίας του ε, ε, με παράνομες διαδικασίες και μέσω κρατικής απόφασης. Είναι μία αρχή η οποία έχει ε, καθιερωθεί από το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη αλλά υπάρχει ένα θέμα αρχής εδώ. Διότι θα σας έλεγα ότι ακόμη κι αν δεν υπάρχει ο χάρτης ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα άλλαζε ε, δεν θα άλλαζε η κατάσταση διότι το άρθρο 51 του χάρτη που περιορίζει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου δεν είναι επινόηση του, χάρτου, του χάρτου απλούστατα περιλήφθη στο χάρτη χάρτη από τη δεκαετία του 60 διότι προηγουμένως δεν σκεφτόμασταν καν να υπάρξει ένας χάρτης ο οποίος υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο όπου είπε ναι ε, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά αρμοδιότης μόνον βάσει του κοινοτικού δικαίου άρα τίποτα δεν αλλάζει. Επίσης, όσον αφορά την εφαρμογή των δύο αρχών του Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων και δικαίωμα εγκατάστασης. Δεν είμαι προσπιστής ε, καμιάς αρχής, αλλά από ό,τι γνωρίζω από την ε, αρχή του, από τις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου δεν βλέπω να υπάρχει ε, κανένα πρόβλημα στην ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων. Η Επιτροπή θα εξετάσει αν ερωτηθεί αν υπάρχει πρόβλημα στην ελεύθερη ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εγκατάσταση των πολιτών, αλλά ε, προημίου δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόσκομα. Παρακαλώ, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει μία αιτιολογημένη απόφαση γραπτός, γιατί νομίζω ότι αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα. Νομίζω ήταν τρία σημεία η το θέμα της Μάριαν Χάρκιν σχετικά με την εγκατάσταση του καταναλωτή, τις αθέμητες μεθόδους και το θέμα που θίξατε σχετικά με τα κεφάλαια. Θα ζητήσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα ζητήματα τα οποία ετέθηκαν σήμερα. Η κυρία Άουκεν. Η Επιτροπή είναι αξιόπιστη και ε, πάντοτε απαντά. Στη Νέα Συνθήκη υπάρχει το άρθρο 2 που αντιστοιχεί στο άρθρο 7 που έχει διάφορα επίπεδα Δηλαδή δεν αναφέρεται ε, μόνο σε ένα θέμα αλλά σε πολλά. Όπως ε, θίξαμε τα θέματα εμείς, οπότε πιστεύω ότι μπορεί κάτι να γίνει. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Κάσμαν ότι έχουμε διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες και ε, ε, δεν πρέπει να ρωτήσουμε την Επιτροπή αν μπορούμε να το πράξουμε, να ρωτήσουμε μεταξύ μας εάν ε, είμαστε σοβαροί και θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε εφόσον έχουμε δυνατότητες να κάνουμε διάφορα. Μία δυνατότητα είναι να θέσουμε μία προφορική ερώτηση προς ζήτηση για το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμόσει τη συστάση που περιλαμβάνει η έκθεση Άουκεν του 2009 οπότε εκεί θα αναφερθούμε στις αθέμητες εμπορικές μεθοδεύσεις και νομίζω ότι ε, οι λύσεις είναι μέσα στην έκθεση Άουκεν. Άρα γιατί να τις ξαναεπινοήσουμε. Ίσως οι συντονιστές μπορούν να σκεφτούν αν μπορεί να γίνει μια προφορική ερώτηση με συζήτηση αντί με ψήφισμα. Ήθελα να στηρίξω με το ε, τελευταίο, δηλαδή να το ελέγξουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών διότι ε, ε, δεν ήμουν τότε μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά τότε αναφερόταν σε θέματα αλληλείας η έκθεση Άουκεν αλλά συμφωνώ να γίνει μία προφορική ερώτηση στο Κοινοβούλιο θα έπρεπε όμως στη συνάντηση συντονιστών να συζητήσουμε επακριβώς το θέμα δηλαδή να δούμε τι αυστηρές επιστολές θα συντάξουμε και θα απευθύνουμε και από ό,τι κατάλαβα από τον συνάδελφο Μάγερ υπάρχουν δύο αρχές, μία η οποία εξέδωσε την οικοδομική άδεια που είπε ότι μπορεί να χτίσεις και η άλλη η Χούντα Νταλουσία η οποία είπε όχι δεν ισχύει και θα κατεδαφίσουμε το οίκημα. Και αυτά είναι θέματα που πρέπει να συζητήσουμε πάλι στη συνεδρίαση συντονιστών αλλά έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις της Κομισιόν σχετικά με το ότι δεν πλήττεται η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων. Σωστά, μπορώ να πάω στην Ισπανία να αγοράσω ένα σπίτι και μέχρι στιγμής είμαστε ε, στην ελεύθερη διακίνηση. Μετά όμως κάποιος μου κατεδαφίζει το σπίτι μου, έχασα τα χρήματά μου, άρα δεν υπάρχει πλέον ελεύθερη ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων. Είμαι σε μία μαύρη τρύπα. Κάπου επένδυσα τα χρήματά μου και κάποιος μου τα πήρε. Ε, διότι θα έπρεπε να μπορώ να τα ξαναβγάλω. Ελεύθερη διακίνηση δεν σημαίνει ότι κάπου βάζω χρήματα και μετά εκεί ε, ε, εξαφανίζονται. Η ελεύθερη διακίνηση σημαίνει είσοδος και έξοδος. Όταν λοιπόν κάποιος καταστρέψει, αφήσει την επένδυσή μου. Δεν είμαι εγώ με νομικός, είμαι απλώς πολιτικός, αλλά δεν τα βλέπω σωστά έτσι. Αν έχουν κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Do you have any... Έχετε κάποιες παρατηρήσεις? Θα ήθελα, δεδομένου ότι είναι σαφές ότι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να δράσει η Επιτροπή σας για το θέμα αυτό είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το θέμα αυτό δεν διέπεται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη και επομένως ε, η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικομάτων δεν εφαρμόζεται σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα να πω τον ε, κύριο που έκανε τα σχόλια ότι δύο ε, βασικοί ένικοι των ε, κατοικών αυτών που αφορούν την ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων και την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει στο Κοινοβούλιο και σε εμά ε, τις αναφέρουσες γιατί θεωρείτε ότι δεν ε, αφορά την Ευρωπαϊκή Συνθήκη το θέμα αυτό. Όσον αφορά το δεύτερο σχόλιο που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι όσοι ε, πλήττονται από την κατάσταση αυτή της κατάχρησης της αστικής δόμησης θα έπρεπε να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού θα έχουν εξαντλήσει όλα τα νομικά ένδικα μέσα στην Ισπανία, ε, είμαι βέβαιη ότι βάσει του ισπανικού νομικού συστήματος μπορεί να χρειαστούν 10 χρόνια μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο. Τα, οι πολλοί από αυτούς που έχουν κατοικίες θα έχουν πεθάνει πριν εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα εντός του συστήματος ε, σε εθνικό επίπεδο. Και όπως ανέφεραν και κάποιοι από τους προελαλήσαντες, εάν κάποιος έχει επαρκή χρήματα και είναι κατά όλων αυτών που προσπαθούμε να επιτύχουμε εμείς, που είναι απλώς να αποδοθεί δικαιοσύνη, τότε μπορείτε κάλλιστα να μας κλειδώσετε στο δικαστικό σύστημα για πάρα πολλά χρόνια. Και πάλι λοιπόν η δικαιοσύνη που καθυστερεί είναι άρνηση δικαιοσύνης ε, για μας. Και επομένως θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θεωρεί ότι αυτό δεν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ε, ε, Έγινε μακροσκελέστατη συζήτηση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών θα συζητήσουμε τη δυνατότητα μιας προφορικής ερώτηση στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό και ε, αναμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντήσεις ε, για τις ερωτήσεις που ήδη ετέθησαν ε, σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ όλους πολύ για τη συζήτηση. Μικρόφωνο παρακαλώ. Να περάσουμε τώρα στην αναφορά του κυρίου Μπέντε Τζούσλακ Γένσεν από τη Δανία σχετικά με παράνομες πράξεις σε σχέση με την κατασκευή ξενοδοχείου στην Εστεπόνα κοντά στη Μάλαγα στην Νότια Ισπανία. Ο κύριος Φλωρίδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη αναφορά αναφέρατε σε ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης στο Δήμο της Εστεπόνα, στη Μάλαγα, ε, στην ε, αυτόνομη περιοχή της Ανδαλουσίας ο αναφέρον αναφέρεται στο σχέδιο κατασκευής ε, παραθεριστικών κατοικιών και ξενοδοχείων στην περιοχή του πρώην ξενοδοχείου Σάντα Μάρτα, κοντά στην περιοχή Ελπαραΐσο Μπαρονάλ, όπου διαμένει. Ο αναφέρον καταγγέλει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ε, με το σχέδιο αυτό, ε, που βρίσκεται πολύ κοντά ε, σε μια πολύ σημαντική παράκτια περιοχή. Ο αναφέρον υπογραμμίζει ότι ε, φιλοξενούνται μοναδικοί οικότοποι και επίσης λέει ότι το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε μια περιοχή μεγάλης οικολογικής σημασίας, υπάρχουν αμόλοφοι στο Μάτας Βέρδες και συμπεραμβάνεται στο δίκτυο δατήρια ε, ε, Natura 2000 και γι' αυτό είναι και σημα, ε, σημαντικής οικολογικής σημασίας. Ε, ο αναφέρον θεωρεί ότι θα υπάρξει πολύ σημαντική ε, υλοτόμηση και θα πληθεί η περιοχή της Κώστα Δεσόλ σε ε, μια έκταση τριών χιλιόμετρων στην περιοχή της Εστεπόνα που έχει μεγάλο οικονομικό ε, πλούτο που έχει πολύ σημαντικά οικοσυστήματα και σημαντική κλωρίδα και πανίδα. Ο αναφέρον ζητά ε, να δει κατά πόσον ε, ε, τηρήθηκαν τα όρια για την αξιολόγηση αντικτύπου, για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέτασαν το θέμα και εξέτασαν και τι γίνεται με βάση το περιβαλλοντικό δίκαιο που ε, εφαρμόζεται και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο σε θέματα της αρμοδιότητός σας και όπως ξέρετε τα θέματα χωροταξικής ε, ε, σημασίας είναι κατά βάση αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εξετάσαμε το περιβαλλοντικό κοινοτικό δίκαιο που ισχύει σε αυτή την περίπτωση και αφενός υπάρχει οδηγία αξιολόγησης ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου για σχέδια και για σχέδια αστικής ανάπτυξης και για σχέδια κατασκευής ε, τουριστικών κατοικιών, τα οποία βρίσκονται στο παράρτημα 2 της Οδηγίας για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Επίσης υπάρχει και η οδηγία για το 2001 για το στρατηγικό σχεδιασμό που θα μπορούσε να ισχύει σε αυτή την περίπτωση που είναι συνήθως χώρος στον οποίο εξετάζονται οι συνέπειες ε, από περιβαλλοντική σκοπιά για τέτοια οικιστικά προγράμματα. Επίσης, ε, πέρα από τις παραβολητικές ε, οδηγίες, έχουμε και τις οδηγίες για τα πτηνά του 97 και την οδηγία για τους οικοτόπους του 92 που ισχύουν μόνο εφόσον το συγκεκριμένο ε, έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, για το δίκτυο Natura 2000. Όταν καθορίσαμε το όλο πλαίσιο της υπόθεσης, υπό το φως των ε, πληροφοριών που συνέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατάσταση συνοπτικά έχει ως εξής. Το Γενικό Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου είναι από το 1994 και εξακολουθεί να ισχύει. Και το 2005 ξεκίνησε μία αναθεώρηση αυτού του σχεδίου Αστικής ανάπτυξης, αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη αναφορά ε, και τη συγκεκριμένη περιοχή, θεωρείται περιοχή στην οποία μπορεί να υπάρξει αστική ανάπτυξη, αλλά περιορίζεται μόνο σε τουριστικές χρήσεις και υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για την οικιστική ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Όσον αφορά το δίκτυο Natura 2000, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος τόπος δεν συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις άλλες περιοχές ε, κοινοτικής σημασίας. Ε, υπάρχει δύο μικροί ποταμοί, Γκουανταλμίνα και Γκουανταλμάνσα, που ανήκουν στο δίκτυο 2000 και είναι κοντά στην περιοχή και ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 από τότε που εγκρίθηκε ο κατάλογος ε, για τα ε, στόπους κοινοτικής σημασίας για τη Μεσόγειο του 2006 και επειδή υπάρχει και το Ελσαλαδίγιο Πούντα Ντεμπάνιος που είναι επίσης τόπος κοινοτικής σημασίας που καθορίστηκε το 2008 ως ε, τμήμα του δικτύου Natura 2000. Όπως γνωρίζετε, το δίκτυο Natura 2000 αυτή τη στιγμή έχει καθοριστεί σε επίγειο επίπεδο, σε χερσαίο επίπεδο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται και με τα κράτη-μέλη προκειμένου να ε, ολοκληρώσουμε και τις θαλάσσιες περιοχές. Ε, οι θαλάσσιοι πόροι λοιπόν που βρίσκονται ενώπιον της περιοχής όπου καταγγέλει ο αναφέρον ότι δεν θα πρέπει να γίνει κατασκευή περιλαμβάνονται σε αυτή τη, στο κοινοτικό σχέδιο. Ωστόσο, η περιοχή δεν περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν οργανώσεις που ζητούν να συμπεριληφθεί στο δίκτυο. Όσον αφορά τώρα την ε, κατάσταση του σχεδίου, βάσει των στοιχείων που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το σχέδιο δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ε, λόγω της γενικότερης ε, οικονομικής κατάστασης και του συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου του συγκεκριμένου Δήμου. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, έχουμε, δεν έχει σχηματίσει ε, άποψη ακόμα οριστική. Θέλουμε να λάβουμε κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες από τις αρμόδιες Ισπανικές Αρχής για να διασφαλίσουμε καταρχάς ε, πώς έχει ακριβώς η κατάσταση του σχεδίου, γιατί δεν έχει ακόμα εγκριθεί αλλά ούτε έχει απορριφθεί. Και επίσης θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μηχανισμοί αξιολόγησης και περιβαλλοντικής προστασίας που προβλέπονται για τις, ε, από την οδηγία για τι αξιολογίε περιβαλλοντικού αντικτύπου και θέλουμε να έχουμε και συγκεκριμένες πληροφορίες από τις Ισπανικές Αρχές για το βαθμό προστασίας που θέλουν να προσδώσουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Επομένω, έτσι έχει η κατάσταση για τη συγκεκριμένη αναφορά προ το παρόν. Ευχαριστώ. Απλώς να ευχαριστήσω για τις πληροφορίες και βάσει των όσων ε, μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να ζητήσω να μην είναι ανοιχτό το ζήτημα. Mrs. Oaken, you wanted to... yes. Κύριε Όκεν, θέλετε το λόγο. Thank for the informations. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πιστεύω είναι σημαντικό η Κομισιόν να έχει σφαιρική άποψη, διότι θυμάμαι υποθέσει στην Ισπανία, είναι εθνικό δίκαιο, είναι περιφερειακό, τι Και μερικέ φορέ ακούω ότι αν δεν είναι υπό εθνική νομοθεσία, τότε δεν εφαρμόζεται κοινοτική νομοθεσία. Ήταν ένα επιχείρημα όταν είχα ένα θέμα στη Μαδρίτη και είχε ε, λεχθεί αυτό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να ε, τηρούμε την ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία και να είμαστε σταθεροί ε, για θέματα Natura 2000. Είναι προσωπική άποψη. Είναι ε, λυπηρό όταν μας έχουν μείνει όμορφες ακτές και βλέπουμε πάλι την ανέγερση ξενοδοχείων. Είναι σαν να οι Ισπανοί να μισούν την ίδια τους τη χώρα. Και Κάνω ό,τι μπορούν να καταστρέψουν την ισπανική φύση. Αλλά ε, δεν απόκειται σε εμά να προστατέψουμε την Ισπανία. Ε, ε, προσωπικά σχόλια είναι αυτά. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι ότι πράγματι λαμβάνεται υπόψη η κοινοτική νομοθεσία. Ευχαριστούμε τις πληροφορίες που πήραμε μέχρι τώρα. Οι Πάντα κάτι λάθος κάνω. σχετικά με σχέδιο κατασκευής φράγματος στον ποταμό Σαμπόρ 1 και σχέδιο κατασκευής υδροελεκτρικού σταθμού στην κοιλάδα Σαμπόρ στην Πορτογαλία. από η κυρία Δεφάρια. Δεφαρία. Δεφαρία. Um, Ευχαριστώ. Η Κομισιόν έχει εξετάσει αρκετέ ανακοινώσει ε, για το φράγμα Σαμπόρ. Θα ήθελα να εστιάσω στο κυριότερο ε, θέμα για τις υπηρεσίες που είναι τα αντισταθμιστικά ε, μέτρα αποζημίωσης, τα οποία τίθενται από τις πορτογαλικές αρχές και τον του προγράμματος. Κάτι σημαντικό είναι ότι η ανέγερση αυτού του φράγματος ακολουθείται από μια επιτροπή όπου συμμετέχουν οι συναφείς αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές, επιστήμονες τοπικών αρχών και μη μικρό, Ε, οι αναφέροντες συμμετέχουν και είναι ενημερωμένοι για τη διαδικασία πλήρως και για την εξέλιξή της. Οι υπηρεσίε τη Κομισιόν παρακολούθησαν αυτή τη διαδικασία με τακτικές επαφέ με τον αναφέροντα. Επίσης έχουμε πρόσβαση στην πλατφόρμα και στα έγγραφα και δύο φορέ το χρόνο ε, λάβαμε πλήρη έκθεση για τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί. Μπορεί να θυμάστε ότι στην αρχή η Κομισιόν δεν ήταν ικανοποιημένη με το πακέτο των μέτρων αποζημίωσης που προτείνονταν από τον προμότερ του προγράμματος και είχαμε υποδείξει ε, που ήταν οι ελλείψεις και τι έπρεπε να γίνει για συγκεκριμένες φυσικές αξίες. Αυτό το πακέτο μέτρων αποζημίωσης συμπληρώθηκε στη συνέχεια και ε, αυτό ακριβώς παρακολουθούμε τώρα. Είχαμε μία συνάντηση στις 28 και 29 Μαρτίου με τις πορτογαλικές αρχές ε, στο θέμα αυτό και ενημερωθήκαμε για την υλοποίηση των μέτρων αποζημίωσης. Πολλά μέτρα παρακολούθησης ήδη υπάρχουν. Οι περισσότεροι περισσότερες τοποθεσίες υλοποίησης έχουν εντοπιστεί σε μια περίμετρο πάνω από 140 χιλιόμετρα γύρω από το χώρο. Ένα από τα θέματα ήταν ότι η Κομισιόν ε, πέστεψε ότι δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν τα μέτρα κοντά ε, στο έργο αλλά σε πιο περιφερειακό επίπεδο αυτό γίνεται. Υπάρχει καθυστέρηση όμως στην υλοποίηση διότι είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία αλλά σημειώνουμε ότι η ε, Επιτροπή ε, έχει ανταποκριθεί στο ρόλο της και παρακολουθεί τη διαδικασία, ζητάει ε, ρυθμίσεις και γι' αυτό ίσως να υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Ένα από τα θέματα που είναι σημαντικό για την Κομισιόν είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα αποσμίωσης θα πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως πριν από την πλήρωση του φράγματος. <clears throat> Αυτό προβλέπεται για τα τέλη του 2013. Μέχρι τότε θα παρακολουθούμε την κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε σχετικές πληροφορίες ε, για την ε, Επιτροπή σας μέχρι να ελέγξουμε αν υπάρχει υλοποίηση των μέτρων ε, πριν το τέλος του 2013. Ευχαριστώ. συνάδελφοι, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Άουκεν, οι Ισπανοί προσπιζόμαστε πάρα πολύ καλά τους φυσικούς μας οικοτόπους και τους φυσικούς μας χώρους με την ισπανική νομοθεσία. Όπως για παράδειγμα την νομοθεσία για, το, για τις ακτές που απαγορεύει την κατασκευή ε, κατοικιών ή την αστική ανάπτυξη κτηρίων σε περιοχές ε, κοντά στην ακτή, οι περιοχές γύρω από τις εκτές περιορίζονται και ελέγχεται ο χώρος από τις πιο σημαντικές οικολογικές οργανώσεις του κόσμου. αν ζητούσαμε από την Ισπανία να διατηρήσουν όλους τους φυσικούς οικοτόπους, ε, όλη τη βιοπικιλότητά της και όλες τις περιοχές ε, σημαντικής προστασίας, νομίζω ότι όταν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχει παραβίαση, δεν θα έπρεπε να μένουν ανοιχτές αναφορές, οι οποίες είναι αβάσιμες και δεν είναι αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει τις αναφορές των πολιτών, για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει παραβίαση ή δεν τηρείται η εφαρμογή του κοινοτικού δοκίου. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η Επιτροπή μας θα πρέπει να μην ασχολείται άλλο με αυτές τις υποθέσεις. Υπάρχει το ισπανικό δικαστικό σύστημα το οποίο συμμορφούται πλήρως με όλες τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εκεί θα πρέπει να επιλύονται αυτά τα ζητήματα. Και επομένως η Επιτροπή μας δεν θα ήταν μετά... Ε, μέσω χειραγωγίας και δημαγωγίας ε, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ από πολίτες οι οποίοι δεν τηρούν οι ίδιοι τους κανόνες και κατασκευάζουν αυθαίρετες κατοικίες σε προστατευόμενες περιοχές και μετά έρχονται εδώ και διαμαρτύρονται για τη ισπανική νομοθεσία που σέβεται την κοινοτική νομοθεσία, κατεδαφίζει τα κτίρια αυτά ή τα κυρίσει αυθαίρετα. Αυτό είναι γεγονός και νομίζω ότι φτάνει, έχει συζητηθεί αρκετές φορές ε, το ζήτημα. Επανειλημμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι δεν έχει καμία σχέση με το κοινοτικό ε, δίκαιο για κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις ακτές, ε, με τους φυσικούς οικοτόπους και κατοικίες αυτές έχουν κατασκευαστεί παράνομα. Και όλα αυτά γίνονται για να προστατευθούν βάσει κοινοτικής νομοθεσίας και περιβαλλοντικών κανόνων οι φυσικοί οικότοποι, το τοπίο, οι περιοχές της υπαίθρου και ούτω η καθεξής της Ισπανίας. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένας να υπερασπίσει την Ισπανία και τους Ισπανούς. Η βιοπικιλότητα της Ισπανίας ε, είναι αντικείμενο προάσπισης της Ισπανικής νομοθεσίας που είναι μία από τις πιο προηγμένε παγκοσμίω σε θέματα περιβαλλοντικών υποχρεωτικής νομοθεσίας. Και επομένως, οι αναφορές οι οποίες δεν έχουν σχέση με ε, με παραβίαση κοινοτικού δικαίου θα πρέπει να παραπέμπονται στο ισπανικό δίκαιο. Ε, ε, please. It's a pity you didn't, you were not here before. Είναι κρίμα που δεν ήσασταν εδώ πριν, γιατί αυτό ήταν το θέμα το οποίο συζητούσαμε και μάλιστα για αρκετή ώρα πάνω από μια ώρα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας εξηγήσω ε, λίγο και καταλήξαμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Αποφάσεις οι οποίες ε, θα συζητηθούν συνεδρίες των συντονιστών. Θα εκτιμούσα λοιπόν ιδιαίτερα να υποβάλλετε, αν υποβάλλετε κάποιο έγγραφο, που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Τόσο μικροφόνο είναι. Oh, to, the new, to the case we are discussing now. So, uh, we do not have any apart from the Commission. Δεν υπάρχει ε, κανείς εδώ, ε, εκτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μείνει ανοιχτό το ζήτημα. I, I we were dealing with the... Νόμιζα ότι συζητούσαμε την πορτογαλική υπόθεση. Και έχω ένα μικρό σχόλιο για την πορτογαλική υπόθεση, ένα σχόλιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ξέρουμε τι συνέβη. Επίσης γνωρίζουμε και πώς ε, αναμίχθηκε στην υπόθεση και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγματικά την παρακολουθούμε πολύ επισταμένα αυτή την υπόθεση Δεν ε, ξεχνάμε λοιπόν, σας έχουμε στον κατάλογο και δεν θα σας ε, ξεχάσουμε. Σίγουρα θα, θα σας θυμόμαστε. Ε, Να περάσουμε τώρα στην αναφορά Κρίς Άντριους Ιρλανδικής Ιθαγενείας σχετικά με σχεδιαζόμενο τεφροτήρα απορριμμάτων στη Χερζόνη Πούλμπερκ στον κόλπο του Δουβλίνου και ε, την ε, ε, αναφορά του Ντάμιεν Κάσιντι εν ονόματι περιβαλλοντολογικής οργάνωσης των περιοχών Ρίγκσεντ, Άριστάουν και Σάντιμάουν σχετικά με τα αναπτυξιακά έργα στον κόλπο του Δουβλίνου, το λιμάνι του Δουβλίνου και τις περιοχές Πούλμπερ, Ρίγκσεντ και Νόρθβαλ το λόγο έχει Επιτροπή. Για την πρώτη αναφορά είχαμε ήδη διάφορες ε, κοινωνίες με την Επιτροπή και πρόκειται για οικοδομικές άδειες ε, οι οποίες είχαν χορηγηθεί και η αναφορά ε, καταφέρεται κατά αυτών των αδειών. Θα ήθελα να σας πω που βρίσκεται η κατάσταση τώρα, αλλά προηγουμένως πρέπει να σας πω ότι εξετάσαμε το θέμα αυτό μέσω του πιλωτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στη συνέχεια βάσει των ε, <clears throat> πληροφοριών που μας έδωσε η Ιρλανδική κυβέρνηση θεωρούμε ότι δεν υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου αλλά κατακρίνουμε την νομοθεσία βάσει της οποίας ε, ε, πετράπει αυτό το σχέδιο κατασκευής διότι χρειαζόταν ε, διαδικασία συνένεσης και ε, περιβαλλοντολογική μελέτη και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενήγαγε την ε, Ιρλανδία ε, είναι η περίπτωση C50 του 2009 και ε, δεν, έχει, δεν είχε ακόμη βγει απόφαση τότε όμως στις 2 Μαρτίου ε, βγήκε και το δικαστήριο δικαίωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεώρησε ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεως είναι παραβίαση και ε, ε, θα πρέπει να αλλάξουν οι διατάξεις κατά τρόπον ώστε να μπορέσει τώρα η νομοθεσία να αλλάξει και θα κοιτάξουμε να το προωθήσουμε. Η περίπτωση αυτή όμως δεν αναφέρεται στην συνένεση και την άδεια που χορηγήθηκε σχετικά με τον αποτεφερωτήρα. Όσον αφορά τώρα το τη δεύτερη αναφορά, η οποία αναφέρεται μόνο στον ε, αποτεφρωτήρα απορριμμάτων, ε, το θέμα είναι παρεμφερές, έχει επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το μόνο επιπρόσθετο ε, που έχουμε να προσθέσουμε είναι ότι απευθυνθήκαμε στη δικαιοσύνη για να έχουμε πρακτικές ε, και αποφασίστη ότι πρακτικές πληροφορίες δεν είχαν δοθεί στο κοινό όσον αφορά τον τρόπο της ε, διεκπαιρέωσης της αποφάσεως μέσω δικαστικής διαδικασίας. Δηλαδή δεν είχε ε, γίνει σεβαστή η αρμόδια οδηγία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση C47 του 2007 και μπορώ να σας πω το 2010 η Ιρλανδία υιοθέτησε νέα νομοθεσία η οποία επιβάλλει την ε, απέτηση να δοθούν πρακτικές πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τις δυνατότητες αναθεώρησης και ε, η ε, αναθεωρητική αρχή στην ε, Ιρλανδία επίσης αναθεωρεί τις αποφάσεις που έχει λάβει άρα εμείς κλείσαμε την παραβίαση σχετικά με το νομικό σκέλος όσον αφορά το άλλο σκέλος δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παραβίαση όσον αφορά την ε, αδειοδότηση, τουλάχιστον όχι μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Προτείνετε δηλαδή να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Τι θέλετε. Υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις δύο αυτές αναφορές τότε τις κλείνουμε. Και η τελική είναι της κυρίας Αγγελικής Χαροκόπου, ελληνικής ηθαγενείας, που εκπροσωπεί 19 ελληνικές οργανώσεις προστασίας των ζώων σχετικά με την εγκύκλιο των ελληνικών αρχών για τη μεταφορά των δέσποτων γατών και τη μη συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτό ο κύριος Φίζελ της Επιτροπής. Γεια σας κύριε κύριοι από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, κύριος Φιούζελ. Αυτή η αναφορά ε, έχει να κάνει με την παρεγκατάσταση των αδέσποτων ε, ζώων συντροφιάς, γατιών και σκυλιών κυρίως ε, και έχει, υπάρχει επίσης και διασυνοριακή μετακίνηση. Το ένα θέμα έχει να κάνει με την Εθνική Νομοθεσία για την ιδιοκτησία ζώων ε, συντροφιάς και το δεύτερο είναι αυτό το θέμα της διασυνοριακής μετακίνησης ζώων συντροφιάς για μη εμπορικούς σκοπούς. Αυτό είναι το μέρος που είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον κανονισμό 998. Υπήρχαν ε, μια-δυο ερωτήσεις ε, σε αυτή την αναφορά σχετικά με την αναγνώριση των ζώων που επιτυγχάνεται με συνήθως με, τοποθέτηση πομπού τσίπ ε, και με διαβατήριο που θα πρέπει να συνοδεύει τα ζώα συντροφιά όταν μετακινούνται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όταν συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή ένα άτομο που ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τους. Το ερώτημα για που, έχει, ε, που αναφέρεται εδώ είναι διτό. Πρώτα, ε, να διασφαλιστεί η μοναδικότητα των μικροτσίπ ε, με τον κώδικα του κατασκευαστή και τον κώδικα της χώρας. Δεν υπάρχει κάτι εναντίον της χρήσης μιας συντομογραφίας για την Ελλάδα στον, στον κωδικό ISA. Όμως αυτό αυτό δεν μπορεί να είναι το μόνο θέμα, διότι οι σκύλοι και γάτες μπορεί να μετακινήθηκαν πριν διασυνοριακά. Ε, πετυχαίνουμε την μοναδικότητα μέσα από τους κωδικούς ISO και το μικροτσίπ σχετίζει το ζώο στο διαβατήριο όπου υπάρχει ή ε, ο εμβολιασμό κατά της λύσα που είναι σημαντικός για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Αυτό είναι ο σκοπός της νομοθεσίας ε, για την οποία συζητάμε τώρα. Υπάρχει ένα άλλο θέμα σχετικά με τον ε, αριθμό των ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την υπάρχει η ελληνική νομοθεσία που περιορίζει την διοκτησία ζών συντροφιάς αλλά αυτό δεν αντανακλάται στην κοινοτική νομοθεσία. Υπάρχει μόνο ένας περιορισμός σε ορισμένους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται εάν είναι πέραν των πέντε ζών που εισάγονται από τρίτες χώρες. Αλλά η κοινοτική νομοθεσία δεν θέτει όριο στην μετακίνηση ζώων συντροφιάς. Δεν ισχύει αυτό εδώ. Η μετακίνηση για μη εμπορικού σκοπούς, όπως φαίνεται και στον κανονισμό 998, δεν έχει την έννοια του μόνιμου ή μη μόνιμου επιστροφή ή μη επιστροφή. Το ζώο μετακινείται διότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να μετακινηθεί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ζώου συντροφιά. Δεν ε, μετακινείται το ζώο για σκοπούς αγώνων, αλλά ακολουθεί, συντροφεύει τον ιδιοκτήτη του. Και συζητούσαμε το πρωί για την ελευθερία διακίνησης ατόμων και αυτά ε, ε, επιτρέπεται να μετακινηθούν, αλλά είναι το άτομο που μετακινείται συνοδευόμενο από το ζώο συντροφιά. Και εδώ δεν ρυθμίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα, για ποιο σκοπό. Δεν είναι όμως για εμπορικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να απολυθεί το ζώο ή να αλλάξει διοκτησία. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία έχω πάρει εντολή να διευκρινίσω σε σχέση με την ε, αναφορά υπό εξέταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, όμως, έξω με ενημερώνει η γραμματεία, θα ήθελα να είναι παρούσα εδώ η αναφέρουσα, αλλά συλλέγει επιπλέον στοιχεία και τεκμηρίωση. Προτείνω λοιπόν να το αφήσουμε ανοιχτό το ζήτημα για κάποια επόμενη συνεδρίαση, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλα γίνονται όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ. Ωραία, συμφωνείτε. Καλώς. Υπάρχει κάποια πρόταση για αναφορές οι οποίες θα κλείσουν από την κατηγορία Β να παραμείνουν ανοιχτές και να ε, συμπεριληφθούν στην κατηγορία Α. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα γιατί ένας από τους αναφέροντες ήταν παρόν, αλλά δεν του ζητήθηκε να... Α, συγγνώμη, ήρθε στην αίθουσα, και δεν ήξερε πού να έρθει. Oh, he's now... What is he going to do if he's now downstairs? Well, we, we can bring him to the room, but shall we reopen the item? I don't know. It's, it Δεν ξέρω τι γίνεται. Αφορά την υπόθεση για το Δουβλίνο και τον αποτεφρωτήρα. Είναι η προηγούμενη αναφορά για τον κόλπο του Δουβλίνου και τον αποτεφρωτήρα. Σας πειράζει να ζητήσουμε από τον ε, αναφέροντα να έρθει, διότι είναι στην είσοδο. Θα μπορούσε να έρθει σε δύο λεπτά. Ας του δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσει. υπάρχει Όλες οι αναφορές ε, στην κατηγορία β' μπορούν να κλείσουν. Ωραία. Oh. Two 27 ε, Υπάρχουν δύο αιτήσει για την 27 και την 93. Ε, Ο κύριος Μποστινάρου ζητά να μεταφερθούν στην κατηγορία Α, οπότε να συζητηθούν. so, what are we doing? Is he coming or not? Is he coming or not? Where from? Έρχεται, από πού έρχεται. Διότι αν έρχεται Πέντε λεπτάκια θα πρέπει να περιμένουμε σίγουρα. Αυτά είναι... Ε, ε, Αυτό τώρα γελίο, μόνο και μόνο να μας χαιρετήσει και να φύγει. Θα μας πει ναι. τώρα για τον ναι, Νταμπέ. Μπορούμε και τα μέλη έχουν φύγει, αλλά ο άνθρωπο έλαβε δηλαδή πρόσκληση και δεν απάντησε ποτέ και τώρα σε εθνικά εμφανίζεται. Αχ, Πόσο που να βγάλαν κάρτα, από τώρα θα βγάλουν κάρτα.